Colleghi, buongiorno. Diamo inizio ai lavori di questa sessione. Ξεκινάμε λοιπόν τις ε, εργασίες μας. Ε, ξεκινάμε με τις ε, ανακοινώσεις από τη συνεδρίαση των συντονιστών. Σήμερα το πρωί αποφασίσαμε να οργανώσουμε την αποστολή στη Μαντρίτη για να ερευνήσουμε το τι ακριβώς έγινε σχετικά με τις ακτές ε, εντοπισμό ακτών στην Ισπανία. Όσον αφορά στα άλλα θέματα της ε, ημερήσεις διάταξης των ε, συντονιστών, νομίζω ότι τις, ε, θέλω να σας πω τις αποφάσεις τις αναβάλλουμε. Θα τις λάβουμε στις επόμενες συνεδριάσεις. Έτσι λοιπόν ε, υπήρξε κάποια συζήτηση ε, με τους συντονιστές σχετικά με τις αποστολές στην Ελλάδα και στην Πολωνία. Και αυτό μετά από πρωτοβουλία του ΕΛΚ σχετικά με τα, το θέμα των υδάτων κατόπιν αρχίσαμε να συζητάμε με περισσότερες λεπτομέρειες το νέο σύστημα επικοινωνίας της Επιτροπής μας με βάση ένα έγγραφο εργασίας ε, το οποίο επεξεργάστηκε η Γραμματεία και επαναλάβαμε ότι είναι απαραίτητο η Επιτροπή αυτή να βρει έναν διαφορετικό τρόπο εργασίας για να αποφύγει τη σόρευση αναφορών. Τώρα, το σχέδιο της ημερήσιας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης της Επιτροπής θα σας διανεμηθεί και τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν στους συντονιστέ, θα υπάρχουν στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την πρώτη ανταλλαγή απόψεων για την ετήσια έκτηση του 2012, η γνωμοδότηση για τη Χάγη, ε, για τη Γαλλική κατόπιν οι ε, αναφορές σε σχέση με την ανικανότητα, ε, με την Ισπανία και με τις Ουγγρικές συντάξεις. Δεν υπάρχουν άλλα θέματα που έχω να σας πω σχετικά με τις ε, αποφάσεις των συντονιστών. Ε, κατόπιν τούτου, περνάμε στο επόμενο θέμα της μερικής διάταξης. Πρόκειται για την έγκριση του σχεδίου μερίσιας διάταξης. Τα βασικότερα θέματα είναι η ψηφοφορία σχετικά με την ε, Ιταλία. Πρόκειται για την διερευνητική μας επίσκεψη για τις ζημιές που έχουν προκληθεί στο περιβάλλον, ε, κυρίως ε, σε περιοχές ε, οι οποίες είναι προστατευμένες. Το 21 στην ημερήσια διάταξη διαγράφηκε γιατί πήραμε μια ανακοίνωση σχετικά με την απόφαση που ελήφθη για αυτήν την αναφορά. Επίσης θέλω να σας πω ότι όσον αφορά στα θέματα 10, 11 και 13 τα ε, θέματα αυτά ε, θα γίνουν παρουσία της αναφέρουσας των αναφέροντων γενικότερα. Επίσης, ε, η ε, αναφορά παριθμών 14, 15, 17 και 19 και 20. Και εκεί θα γίνει, θα υπάρχει παρουσία των αναφερόντων. Το 23. Επίσης και εκεί θα έχουμε αναφορά ε, εξ ονόματος της Άρκα Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην πολύ σημαντική ακρόαση η οποία έλαβε χώρα εχθές, ακρόαση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Μία ακρόαση την οποία οργανώσαμε μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τις Επιτροπές ε, Λίμπε και Γιούρι. Και ε, θα ήθελα να ευχαριστώ κυρίως ε, τη Γραμματεία για τη δουλειά που έκανε σχετικά με την ακρόαση αυτή για να καταστεί δυνατόν η ακρόαση να λάβει χώρα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο συνάδελφος Τουργκάης ζήτησε το λόγο. Όχι, δεν αφορά αυτό το σημείο, κύριε Πρόεδρε. Σας άφησα να τελειώσετε γιατί Μα είπατε για αυτές τις ε, ανακοινώσει και για τι αποφάσει των συντονιστών. Αυτό που θέλω να πω είναι ένα ζήτημα το οποίο το είχαμε στην ημερήσια διάταξη για τη 1266 ε, αναφορά θέλω να σας πω που υπήρχε και είπαμε να ξανά ανοίξει. Οπότε εμείς δεν συμφωνούμε γιατί δύο φορές έχει ξανασυζητηθεί αυτή η αναφορά Πρόκειται για ένα κλίβανο, ε, ε, μια από αποτέφρους τέλος πάντων. Λοιπόν, συζητήθηκε, έκλεισε, ξανασυζητήθηκε, ξανάκλεισε. Δεν έχουμε καινούργια στοιχεία. Γι' αυτό σας λέω διότι, ότι εδώ πέρα δεν υπάρχει λόγος για τρίτη φορά να επανέλθει το ίδιο θέμα. Γι' αυτό σας λέμε. Να μην ξανανοίξει αυτή η αναφορά. 1266-2009. Ε, está aquí. 1266. βεβαια είναι μια πρόταση για την οποία δεν προβλέπεται ψηφοφορία. με πάση περιπτώσει, εμείς θα λάβουμε υπόψη μας ε, όλα αυτά που ελέγχθησαν σχετικά με την αναφορά αυτή του 2009. Οπότε, Αφού είναι έτσι, να το ζητήσουν τουλάχιστον οι συντονιστέ. Γιατί στα έγγραφα τα οποία μοιράσατε έχει ε, αναφερθεί αυτή η αναφορά. Εμείς θέλουμε να κλείσει. Επειδή λοιπόν υπάρχει βέβαια αυτή η αναφορά με τις ε, αντιρρήσεις του κυρίου Τουρκάης, ε, δεν θα αποφασίσουμε, δεν θα ξανανοίξουμε αυτή την αναφορά. Πολύ ωραία. Άρα δηλαδή δεν μπαίνει στις αναφορές που θα ξανασυζητηθούν. Συνάδελφος Κολάσκα. Να σας ρωτήσω, να ζητήσω κάτι για την ε, ψηφοφορία. Quindi approvata l'agenda di oggi. Κοιτάξτε, εγκρίθηκε η σημερινή ημερήσια διάταξη. Δεν βλέπω να υπάρχουν άλλες αντιρρήσεις για την σημερινή ημερήσια διάταξη. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Sí, señora Presidenta. Ναι, en este punto eh, eh, en la medida en que hay un tema. Θέλω να σας πω, διότι εδώ πέρα υπάρχει θέμα αρμοδιωτός μας. Είχε γίνει ανταλλαγή ανακοινώσεων και επικοινωνιών εντάξει ημών και εμού και με τη γραμματεία. Είχαμε εδώ πέρα δύο Ισπάνους. Δύο Ισπάνους. Πρόκειται για τον αναφορά 1201 και 1209. Δεν οι δύο αναφορές αφορούν κάποια βρέφη, τα οποία εκλάπησαν στην Ισπανία μεταξύ 1950 και 1990. Είναι θέμα το οποίο απασχολεί χιλιάδες Ισπανών και έχει να κάνει με τα ανθρώπινα δικαιώματα και πώς θα αντιλαμβανόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό θεωρώ ότι αυτές οι αναφορές αξίζει να ζητηθούν στην Επιτροπή μας. Άρα θα πρέπει να γίνει σχετική διόρθωση στα έγγραφά μας και θα πρέπει όμως να εξεταστεί από την Επιτροπή μας αυτή η αναφορά. Γιατί έχουμε το συγκεκριμένο πρόσωπο στη συγκεκριμένη αναφορά, αλλά θα πρέπει να το γενικεύσουν το ζήτημα. Και οπότε θα πρέπει επομένως να ακούσουμε αυτούς που επιζήτησαν να ακουστούν ε, μέσω αυτής της ε, αναφοράς. Grazie collega, abbiamo preso in considerazione i suoi rilievi. Πολύ ωραία, θα λάβουμε υπόψη μας ε, τις δικές σας απόψεις και έχει αλλάξει αυτή η αναφορά, πλέον ε, έχει γίνει αποδεκτή και αυτό το θέμα θα το επισημάνω ε, στις συνεδρίες των συντονιστών την επόμενη φορά. Πάμε τώρα στο σημείο υπαριθμών 3 της ημερήσιας ε, διάταξης, έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων 6 Νοεμβρίου και 3 Δεκεμβρίου. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνονται αυτά τα πρακτικά. Δεν βλέπω να υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνονται λοιπόν τα πρακτικά. Δεν υπάρχουν άλλες ανακοινώσεις, ούτε έχει ζητήσει κανείς το λόγο. Περνάμε στο σημείο υπερτιμών 7 τη ημερήσια διάταξη, ε, που είναι η ψηφοφορία σχετικά με την έκθεση ε, που αφορά στη διερευνητική επίσκεψη στην Ιταλία. Συνάδελφος Μέρκες, θέλετε να λάβετε το λόγο μετά. Κατόπιν τούτου μπορούμε να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Η γραμματεία μου λέει ότι οι πράσινοι είναι τέσσερις, αλλά κατ' ουσίαν οι τρεις έχουν δικαίωμα ψήφου. Αυτό το είπα γιατί μου το ζήτησε να το πω επιτροπή. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ψηφίζουμε. Τροπολογία 1 για τη σύσταση 1. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική, ηλεκτρονικός έλεγχος, επαλήθευση. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Να κλείσουμε την ψηφοφορία. Έκλεισε λοιπόν η ψηφοφορία. Δεκατέσσερις υπέρ, 12 κατά, εγκρίνεται η τροπολογία. Τροπολογία 2 για τη σύσταση 2. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Υπέρ, κατά, αποχές, Ελεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίφθηκε η τροπολογία. Πάμε στην τροπολογία υπαριθμών 3 για τη σύσταση υπαριθμών 4. Υπέρ παρακαλώ. ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Το ίδιο αποτέλεσμα απορρίπτεται. Πάμε στην ε, υπαριθμών 5 για την ε, συν 4 για τη σύσταση 5 ψηφίζουμε. Τροπολογία 4, σύσταση 5, έκλειση ψηφοφορία. Ψηφίσαμε για την τροπολογία 4, σύσταση υπαριθμών 5. Ψηφίζουμε λοιπόν. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται 14 υπέρ, 11 κατά. Τροπολογία 5, σύσταση 8. Ζητήθηκε ψηφοφορία σε τμήματα. Ψηφίζουμε για το πρώτο τμήμα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές θα έλεγα να επαληθεύσουμε για το δεύτερο τμήμα της ε, τροπολογίας 5. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται η τροπολογία. Πάμε στην τροπολογία 6, ε, σύσταση 8, υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία τεχνική η 7 για τη σύσταση 8α, υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για το σύνολο της έκθεσης. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Ομόφωνα. 27 υπέρ. Ε, συγχαίρουμε τη συνάδελφο Μέργκες και της δίνω το λόγο για να σχολιάσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αναφέροντες. Γιατί για ένα τέτοιο μόνιμο πρόβλημα στην Ιταλία είχαν το θάρρος να βγουν μπροστά και να θελήσουν να ακουστούν. Ακούστηκαν. Είναι πολύ σημαντικά τόσα καταγγέλουν και είναι πάρα πολύ σημαντικό να συζητήσουμε αυτά τα οποία καταγγέλουν στην Επιτροπή των Αναφορών. Και θα πρέπει έτσι να αποδείξουμε ότι οι πολίτες μπορούν να αλλάξουν το, το, περιβάλλον τους και στη χώρα τους και στη, στην Ευρώπη. Κάθε ψήφος μετράει, οπότε θα ήθελα κι εγώ να ευχαριστήσω τους συναδέλφους οι οποίοι ε, κάνουν ό,τι μπορούσαν και οι αναπληρωτέ, τα, τα, τακτικά μέλη, όλοι αυτοί οι οποίοι στην ερευνητική των πραγμάτων επιτροπή συμμετέσχουν, όλοι μαζί επομένω, ε, χέρι-χέρι δουλέψαμε και αν δείξουμε επομένω ότι είμαστε πάντα έτσι σημαίνει ότι διακομματικά μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και νομίζω ότι θα πρέπει όλοι οι Ιταλοί πολιτικοί να συνεργαστούν για αυτό το πρόβλημα, γιατί πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο ε, έχει πάρει δεκαετίε Και γι' αυτό θα πρέπει να επιληθεί ακόμα και μέσα στη συγκυρία τη κρίση. Πρόκειται για μια ευκαιρία που έχουμε τώρα. Ε, και θα πρέπει να δούμε επομένω τι θα γίνει με τι Ιταλικέ εκλογέ που δίνει το Σαββατοκύριακο και ε, πιστεύω ότι δεν υπάρχει πολιτικός ο οποίος δεν θα δεσμευτεί να κάνει κάτι στη νέα εντολή, στη νέα θητεία τέλο πάντων. Επίσης ευχαριστώ την ε, γραμματεία που βοήθησε τόσο πολύ, ώστε να πετύχει αυτή η ερευνητική επιτροπή, η ερευνητική αποστολή και νομίζω ότι την επόμενη φορά που θα πάμε Ιταλία να μην έχουμε το πρόβλημα αυτό με τα σκουπίδια και μια που είμαστε στον 21ο αιώνα αντιμετωπίζουμε τα σκουπίδια σαν, μια, σαν ένα πόρο και όχι σαν ε, κάτι άχρηστο. Ευχαριστούμε. Με κυρία Και δίνει το λόγο στην κυρία Άουκιν. Εγώ θέλω να έρθω και να συμφωνήσω με αυτά. Συμμετέχουν στην αντιπροσωπεία και νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καλή η συνεργασία μας. μπορέσαμε να ε, ωφεληθούμε από την εμπειρία όλων. Ήταν υπέροχη η δουλειά της Επιτροπής αυτής. Και νομίζω ότι διαπιστώθηκε το ότι πετύχαμε πολλά και Ελπίζω να μην ξαναπάμε σύντομα για το ίδιο πρόβλημα, αλλά πάντω όταν ξαναπάμε πιστεύω ότι θα διαπιστώσουμε ότι η Ιταλία ε, και αυτή θα, θα βοηθήσει στην ε, νέα κατάσταση των πραγμάτων και τα σκουπίδια και νομίζω ότι εάν μπορέσουμε να κάνουμε να ισχύουν όλα αυτά τα οποία έχει θεσπίσει σαν η Ευρωπαϊκή Ένωση τότε θα έχουμε 420.000 θέσεις απασχόλησης. Αυτό δεν θα πρέπει ποτέ να φεύγει από το μυαλό μας η διαχείριση του των απορριμμάτων αφορά και αυτή την πτυχή. Ούτε γίνεται υπεργολαβία με τέτοιου είδου θέσει απασχόληση. Να, ένα πάρα πολύ έξυπνο τρόπο να βοηθήσουμε να βρεθεί διέξοδο από την κρίση. Βεβαίω θα πρέπει να ευχαριστούμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολύ ωραία. Κυρία Όκεν, από ό,τι βλέπω κανείς άλλο δεν ζητάει το λόγο. Πάμε στο επόμενο σημείο της σημερινή διάταξη, που είναι ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την ε, διερευνητική επίσκεψη στη Γαλλικία. Ο συνάδελφο κύριος Μπουλόν έχει το λόγο που ε, ήταν και ο επικεφαλή ο αρχηγό τη αποστολή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε πάει στην Γαλλικία για αυτή την, την αποστολή. Οπότε, όπως θα πούν και οι τα πήγαν πάρα πολύ καλά. Αγαστή συνεργασία. Όλοι, όλοι, πληρωτές, τακτικοί όλοι. τοπικές αρχές, ε, είδαμε, τους αναφέροντας είδαμε και διαπιστώθηκε ότι ήταν βάσιμο τόσο καταγγέλλοντα. Βέβαια, ήταν μια διαδρομή 15 ετών. Πάντως πήγαμε με τοπικέ αρχέ και με τους και ε, επισκεφθήκαμε πολλούς αυτούς τους κόλπους της Γαλλικής, αυτά τα φιόρδε τέλο πάντων, τα ρία τα λένε. Είδαμε και κάποιες άλλε εγκαταστάσεις που ήταν κοντά σε, ε, σε αστικές περιοχές, για ε, πετροχημικές εγκαταστάσεις ε, κοντά σε, στη φύση, σε πολλές ε, περιπτώσεις τα προβλήματα είχαν επιληθεί. Αλλά πάντως εμείς πήγαμε εκεί που καθαρίζονται τα ύδατα και τέλος πάντων είχαν διαπιστωθεί κάποιες παραβιάσεις από πλευρά Ισπανίας, τοπικές αρχές κάνουν μεγάλη προσπάθεια, ε, πήγε καλά η συνεργασία μας, κατεβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια και από ό,τι φαίνεται, λέω από ό,τι φαίνεται γιατί εμείς δεν μπορούσαμε να διαπιστώσουμε 100% τι γίνεται, από ό,τι φαίνεται λοιπόν τώρα τηρείται η οδηγία για τα ύδατα. Καμιά φορά κάνουμε και περισσότερα από όσα απαιτεί η οδηγία. έχουν φτιάξει ένα σωρό εγκαταστάσεις καθαρισμού των υδάτων και στο Φερόλ και στο Βίγκο. Δεν μας έκρυψαν οι τοπικέ αρχές ότι ακόμα υπήρχαν κάποια πράγματα προς βελτίωση. Το σύστημα ακόμα επιδέχεται βελτιώσεις. Και σε τελευταία ε, κόλπο που σκεφτήκαμε είδαμε ότι υπάρχουν εκεί κάποιες λάσπες, ε, οργανική ύλη ε, που φτάνει τα δύο μέτρα σε ύψος και τα τρία τέταρτα του εκεί ποταμού έχουν καλυφθεί από αυτή την ε, λάσπη. Βέβαια υπάρχει μια αστική περιοχή εκεί, υπάρχει χωροταξία καλή με, με πάρκα, με δέντρα Οπότε ακριβώς γι' αυτό ήταν ένα σοκ να δούμε σε αυτή την περιοχή που έχει τόσο ωραίες παραλίες, τόσο ωραίο περιβάλλον, να βλέπουμε τέτοιου είδους ε, απόβλητα, τέτοιου είδους ε, βρωμιές ε, που να είναι εκεί τόσο καιρό. Και είπαν οι τοπικές αρχές ότι προσπαθήσαν εκεί να, να τηρήσουν την οδηγία για τον καθαρισμό. Πάντως το θέμα είναι να δουλέψουμε περισσότερο και εις βάθος, επί τη βάση των στοιχείων, των εγγράφων που έχουμε, για να δούμε αν όντω ε, γίνεται ο καθαρισμός όπως πρέπει και να δούμε τι θα γίνει με αυτή την οργανική λάσπη το, του ύψους των δύο μέτρων ή του βάθους των δύο μέτρων ή του βάθους των δυο μέτρων. Οπότε να δούμε πώς θα γίνει για την κήτη του ποταμού, μια που υπάρχουν ε, κάποιες εταιρείε ε, του αλληλευτικού κλάδου που ασχολούνται με με, τις σπεσιαλιτέ της, τα θαλάσσιες της Γαλλικίας, τα, τα, τα μαλάκια, τα θαλασσινά, που θίγονται και, και αυτές οι εταιρείε. Συναντήσαμε ψαράδες και μας είπαν ότι έχει συρρυκνωθεί πολύ δραστηριότητά τους. Τους έχει χτυπήσει η ανεργία. Κλείσανε ένα σωρό επιχειρήσεις αλληλευτικές. Και η ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν αντιστάθμιση ε, αυτή τη σύγχρονη δραστηριότητα. Ε, Μα οδηγήσει να σκεφτούμε ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι περιφερειακέ αρχέ επίση θα πρέπει να φροντίσουν, τόσο ώστε ο κλάδο ο να σταματήσει να θίγεται, να πλήσεται τόσο πολύ. Αυτά είναι Και επομένως ήταν ε, ενδιαφέρουσα, ήταν ε, αποδοτική αυτή η αποστολή. Ό,τι ρωτήσαμε μας το απήντησαν οι αρχές της Γαλλικής και γι' αυτό σας λέω ότι ήταν ε, τέλεια υποδειγματική συνεργασία μας και ε, βέβαια εμείς θα πρέπει να το ψάξουμε ακόμη περισσότερο να δούμε Και μπορούμε ακόμα περισσότερο να τους βοηθήσουμε για να βελτιωθεί η κατάσταση. Κυρίω όσον αφορά αυτή του την, τη λάσπη που μας σοκάρισε με όλους αυτούς τους αναφέροντες. Και α πούμε παραδείγμα κάποιου γιατί συναντήσαμε και μιλήσαμε ε, και με κάποιου οι οποίοι δεν ήταν στη λίστα των ε, αναφερόντων, αλλά δεν μπορούσαμε να του πούμε όχι μια που ήμασταν εκεί πέρα. Εκεί και βλέπαμε τα μάτια μας τα, τα προβλήματά τους, τα, το δράμα τους, τι είχε υπάρχει το περιβάλλον, οπότε επρόκειται λοιπόν για, για αυτούς του, του, τους άτυπους συνομιλητές μας. Αυτά για την αποστολή μας και ελπίζω ότι συμφωνούν και οι συνάδελφοι που συμμετέσχουν. Α, ας λάβω το λόγο να σας τα πούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπουλάν. Η συνάδελφος κυρία Τσανόκα ζήτησε το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Very... Ελπίζω όντως, να ήταν αποτελεσματική αυτή η αποστολή και θα ήθελα να συγχαρώ τη Γραμματεία και ιδιαίτερα την Ιβέτ και τον Δαβίδ που συνέβαλαν τόσο πολύ στην διοργάνωση της επίσκεψης αυτής. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, επισκεφθήκαμε τρεις πόλεις, μιλήσαμε με δεκάδες αναφερόντων και Βγάλαμε και τα πρώτα συμπεράσματα που παρουσιάσαμε στην προηγούμενη συνέντευξη τύπου μας. Ότι δηλαδή έχουν βάση αυτές οι αναφορές. Με βάση αυτά που μας είπε ο κύριος Μπολάν, συναντηθήκαμε ανεπίσημα και με αναφέροντες και αναφέρουσες που, τον οποίων οι αναφορές δεν είχαν ακόμη εξεταστεί στην Επιτροπή μας, γιατί υπάρχουν ακόμη εκρεμή προβλήματα. Επισκεφθήκαμε τρία δέλτα ποταμών και Είδαμε πού υπάρχουν τα περισσότερα προβλήματα. Αλλά οι εκπρόσωποι των αρχών μας είπαν ότι η ποιότητα των υδάτων είναι μέτρια. και ότι βρίσκουν στο είδωρ πολλές ουσίες. Ουσίες, το λέω για να μην πω τίποτα χειρότερο. Και πρέπει να καθαρίζεται τακτικά σε βάθος μέχρι και δύο μέτρα. Μέτρα. Βέβαια όλα αυτά συμφωνούν οι πολιτικές ομάδες ότι θα δημιουργήσουν ε, θέσεις εργασίας και μάλιστα πράσινες ο καθαρισμός των υδάτων δηλαδή. Αλλά ακούσαμε και εμπειρογνώμονες, που είχαμε μαζί μας δηλαδή, αλλά δεν εξετίμησα ιδιαίτερο στο γεγονός ότι οι αρχές δεν μας απάντησαν για τις επαφές τους με τους αναφέροντες. Γιατί η πρώτη σχετική αναφορά είναι του 99 μετά 2006-2007 και ούτω καθεξής. Καθ' όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν οι αρχές, κάτε με, οι αρχές λέγω, από ό,τι κατάλαβα από τις παρουσιάσεις που μας έκαναν, δεν συνήψαν σχέσεις με τους αναφέροντες. Μίλησαν για κάτι στο σελίδες όπου μπορούν να πάνε οι αναφέροντες να βλέπουν πληροφορίες, αλλά δεν είναι αυτός ο σωστός τρόπος εργασίας, αλλά η προσωπική επαφή. τι φοβούνται αυτές γιατί καμιά φορά λένε ότι είναι εκνευρισμένοι οι αναφέροντες όταν βλέπουν τις αρχές. Αλλά είναι κάτι αναπόφευκτο. Αυτό ήταν το πρώτο συμπέρασμα από την επίσκεψή μας, ότι πρέπει να βελτιωθούν οι σχέσεις των Υπουργών και άλλων αρχών με τους αναφέροντες για να λυθούν αυτά τα προβλήματα που διαπιστώσαμε. Άρα, να, αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε ο κύριος Σάντσεφ Πρεσέδο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θεώρησα ότι η αποστολή στη Γαλλικία ήταν πολύ καλή. Η... Τα μέλη της αντιπροσωπείας και η πρόεδρος τα έκαναν όλα πολύ καλά και το αποτέλεσμα νομίζω επίσης είναι πολύ καλό. Είχαμε παφάς με τους αναφέροντες και μπορέσαμε να δούμε τα πράγματα με τα μάτια μας. Και οι ίδιοι ενδιαφερόμενοι δέχτηκαν ότι ήταν θετική η επίσκεψη, είχαμε επαφές και με τις αρχές, βεβαίως. Αρχές. Δεν είχαμε βέβαια επίσημη πρόσκληση από όλες τις αρχές, δεν ήρθαν όλες οι αρμόδιες αρχές να αντιπροσωπευτούν εκεί και αυτό ήταν κρίμα, αλλά είδαμε τουλάχιστον επιτοπίως τα πράγματα. Καλύψαμε δηλαδή το θέμα και των σχέσεων με τους αναφέροντες που έχουν έρθει εδώ στην Επιτροπή μας αλλά που δεν έχει διεκπαιρεωθεί ακόμα η αναφορά τους και έτσι τους δείξαμε ότι είμαστε πολύ κοντά στους πολίτες. Εγώ ήμουν μέλος κάποτε της Περιφερειακής Αρχής στη Γαλλικία και ήθελα να δω πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα από τότε. Και αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η ποιότης των υδάτων, η οδησιατική οδηγία δηλαδή που εγκρίθηκε το 2000, δεν έχει συμπληρωθεί ακόμα ε, στην πράξη μέχρι το 2013 που βρισκόμαστε. Υπάρχει λοιπόν καθυστέρηση στην επίτευξη των στόχων. Χρειάζονται φυσικά και πολλές επενδύσεις γιατί η μονάδα καθαρισμού που κατασκευάστηκε έχει τελικά πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες από ό,τι αρχικά είχε προβλεφθεί και όταν θα έχουμε τα χρήματα θα συμπληρωθούν και τα έργα. Στο Ισοφερόλ είδαμε ότι υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη καθυστέρηση και θα έπρεπε να θεωρηθεί προτεραιότητα η συμπλήρωσή τους λόγω της κατάστασης των υδάτων του ποταμού εκεί. Και είναι επομένως πιο δύσκολο εκεί να επιτευχθεί ο στόχος. Και στην Κορούνια είδαμε ότι είχαν προχωρήσει πολύ τα έργα, σχεδόν συμπληρωθεί, αλλά υπάρχουν ακόμα δυσκολίες. γιατί η λάσπη που έχει συσσωρευτεί είναι πολύ ψηλή. Εδώ και χρόνια έχουν γίνει έλεγχοι της ποιότητας των νερού εκεί. Πολύ λεπτομερής έλεγχη των αυτόνομων τοπικών αρχών, αλλά πρέπει ακόμα να γίνουν πολλά για να έχουμε καλή ποιότητα ενωσιακών προτύπων του νερού. Θα δούμε τι θα αναφέρει η τελική μελέτη και αναφορά. Ευχαριστούμε. Μιράντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα αρχίσω ευχαριστώντας την Επιτροπή μας για όσα έχει κάνει και την Πρόεδρο ιδιαίτερα είναι πραγματικά κοινοβουλευτική αποστολή γιατί η Επιτροπή Αναφορών έχει αποδείξει ότι ακούει τους πολίτες. Μερικές φορές στους δύσκολους καιρούς που ζούμε οι κυβερνήσεις δεν δίνουν τη δέουσα προσοχή στις αναφορές. Υπάρχουν μερικές που χρονίζουν και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών που μπορεί να έχουν υπογράψει αναφορά με 5.000 υπογραφές δεν εισακούονται στην Κορούνια, στο Φερόλ, στο Φίγκο. Ορισμένοι μας είπαν ότι δεν υπάρχει επαρκής πληροφόρηση, διαφάνεια και διάλογος με τις τοπικές αρχές. Η αποστολή λοιπόν αυτή έδειξε την ανάγκη που υπάρχει για διάλογο και αυτό ήταν νομίζω θετικό. Επίσης, είναι καλό ότι έγινε δεκτή αυτή η έννοια της ανάγκης καθαρισμού των θαλασσίων υδάτων που εισραίουν σε ποταμούς. Όλοι κατάλαβαν από την αποστολή πόσο σημαντικό είναι αυτό το φαινόμενο που λέμε στα ισπανικά ρία. Είναι θέμα περιβάλλοντος, είναι θέμα υπαίθρου βιοπικιλότητος. Είναι λοιπόν κάτι που αφορά και την καθημερινή μας ζωή στην περιφέρειά μας και αφορά και τις θέσεις απασχόλησης βεβαίως. Ακούσαμε λοιπόν τους αναφέροντες και τις αναφέρουσες που ασχολούνται με υδατοκαλλιέργειες. Πολλοί από αυτούς δεν είναι σε θέση να εργαστούν γιατί δεν υπάρχει, γιατί υπάρχει μεγάλη μόλυνση και ζητούν κάτι να γίνει. Από τους αριθμούς που μας έδωσαν οι τοπικές αρχές όμως είχαμε μια διαφορετική εικόνα. Δεν υπάρχουν διαρθρωτικά, ποσά από τα διαρθρωτικά ταμεία για τη Γαλλικία. Για το σκοπό αυτό ενώ πρέπει τα ενωσιακά κονδύλια να χρησιμοποιούνται πράγματι για το στόχο για τον οποίο διατίθενται. Το, κείμενο, το πρώτο σχετικό κείμενο εγκρίθηκε το 2000. Βέβαια δεν είναι ποτέ αργά, αλλά δεν χρειάζεται και για άχρηστες καθυστερήσεις. Η έκθεσή μας τελικά νομίζω ότι πρέπει να βοηθήσει την επίτευξη αυτών των στόχων την αφαλάτωση ιδιαίτερα, γιατί αν καθαριστούν τα νερά θα αυξηθούν οι θέσεις εργασίας. Για μας είναι όλα αυτά πολύ σημαντικά. Αυτά τα ρίας λοιπόν είναι για μας ιδιαίτερα σημαντική βιότοποι και θέλω να ξαναευχαριστήσω την Επιτροπή μας ολόκληρη, όχι μόνο τα τρία μέλη που πήγαν εκεί, για όλα όσα έχουν κάνει για να ακουστεί η φωνή των πολιτών. Ε, έτσι αυξήθηκε και η αξιοπρέπεια και η αξιοπιστία του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αυτή η επίσκεψη στη Γαλλικία ήταν ε, πολύ ουσιαστική. Βέβαια, ε, θα ήθελα να διαφοροποιήσω λιγάκι τις δύο μέρες. Την πρώτη μέρα στην Βίγκο και τη δεύτερη στη Φερόλ και στην Κορούνια. Το πρωί Πήγαμε στη Φερόλ, αργότερα στην Κορούνια και πρέπει να πω ότι το πρόγραμμα ήταν πολύ φορτωμένο. με ε, πολλές συναντήσεις, ε, πολύ πυκνό πρόγραμμα. Πάντως θέλω να επισημάνω ότι υπήρχε πάρα πολύ καλή συνεργασία των περιφερειακών αρχών. Επίσης, ε, Εκείνο που μας ε, έλειψε, θέλω να πω, ήταν οι θεσμικές ε, επαφές. Δηλαδή, τελικά δεν μπορέσαμε να ε, μιλήσουμε με κανέναν δήμαρχο σε καμία πόλη και η επαφή με τις περιφερειακές αρχές τη δεύτερη μέρα και αυτή ήταν πολύ περιορισμένη. Νομίζω λοιπόν ότι γενικά στην Ισπανία υπάρχει έλλειψη επαφών ανάμεσα στις περιφερειακές αρχές και τους πολίτες. Πάντως αυτή η έλλειψη διαφάνειας με τις περιφερειακές αρχές κατά την άποψή μου αυτό δεν είναι σωστό. Και θεωρούν επομένω και ο κόσμος και οι αρχές ότι είναι αυτό μια προτεραιότητα και όχι μόνο για λόγους υγείας, πρόκειται ε, για το Σαντιάγο που είναι αυτός ο καθεδρικός. Δηλαδή, είναι κάτι πολύ βασικό. Είναι, είναι, είναι η ζωή, είναι η υγεία για την καλλικία, ε, για οικονομικούς λόγους, για, για λόγους τουρισμού. Και γι' αυτό λέμε ότι πρόκειται για μια τεράστια πρόκληση που έχουν λάβει οι Θεσσαριές για να μπορούσαν να είναι στο ύψος των περιστάσεων και να γίνεται αυτό το οποίο ορίζουν οι κοινωτικές οδηγίες. Τώρα κάτι στο οποίο θέλω να επανέλθω. Το λέμε εδώ, το, το, το λέει και αναφορά. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε ότι αυτό που έγινε στη, στη ιστορία αυτού του Μπούργου είναι κάτι το απαράδεκτο. Και θα θυμάστε ότι αυτό που θέλαμε ε, πρόκειται για κάποιο σκάφος το οποίο το είχαν οι αναφέροντες και λέγανε ότι ήταν απαράδεκτο να, να, να πηγαίνουν, να ανεβαίνουν στο σκάφος και να ελέγχουν οι, οι αρχές. Αλλά πήγαμε και συναντήσαμε όλες τις πλευρές και νομίζω ότι δεν θα έπρεπε η Επιτροπή να αποδεχθεί και αυτή την κατάσταση που είχε επιβληθεί και ακριβώς ε, την ίδια μέρα ε, τελικά μπορέσαμε να δούμε τις αρχές και τελικά ε, πιεζόμασταν από τον χρόνο, δεν μας είπαν αρκετά. Δεν υπήρξε ισορροπημένη κατανομή του χρόνου. ήτανε υπήρχε μια, κάποια μονομέρεια και τώρα ολοκληρώνω. Τα τελευταία 20 χρόνια στην Γαλλικία ε, γιατί χρειάζεται να βλέπουμε κάποιον προοπτική εμεί οι πολιτικοί τα πράγματα. Υπήρχαν κάποιε πολύ θετικέ εξελίξει, γίνανε τεράστιε προσπάθειε το 89. Είχαμε μόνο μία εγκατάσταση καθαρισμού των υδάτων. Για, ήταν, δηλαδή καθαρισμό ε, για 10.000. Τώρα έχουμε 150-150 για, για 3 εκατομμύρια κατοίκου. 150 τόσε λοιπόν εγκαταστάσει για 3 εκατομμύρια. Βλέπετε επομένω ότι συνεχίζει για η αρχή του τόπου να εκτελεί τις ε, κοινοτικές οδηγίες, να ε, κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν στα ρίας, εκεί στα, στα ποτάμια, στα, στα, στα φιόρδ, ε, στο, στο φερόλ και είδατε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για να λυθούν αυτά τα προβλήματα της περιφέρειας και των πολιτών. Σας ευχαριστούμε κύριε Μιγιάν. Ε, το λόγο έχει ο κύριος Μάγερ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ τώρα να συνεχίσω τα, τα, τα, τα συγχαρητήρια ε, της, ε, προς, προς την αντιπροσωπεία μας, προς την ε, ε αποστολή όπως, που ήταν υπηρεσίας ο κύριος Μπελάν. και νομίζω ότι έτσι φαίνεται το πόσο αντιποκρινόμαστε στον κόσμο που απευθύνεται σε εμά και από την άλλη μεριά ο κόσμος αισθάνεται αγανακτισμένος, αγανακτή κατά των αρχών οι οποίοι δεν θέλουν να δεσμευτούν, να πούνε συγκεκριμένα πράγματα. Πότε θα κάνουν αυτό το οποίο πρέπει για να καθαρίσουν τα, τα, τα, τα ποτάμια, τα ποτάμια και τις θάλασσες. Επιβάλλεται να το κάνουν και δεν το κάνουν. Μιλάμε τώρα για διαδρομή 13-15 ετών και γι' αυτό είναι λογικό να αγανακτεί ο κόσμος. Και αυτή η αγανάκτηση θα πρέπει επομένω να γίνει μια θετική προσπάθεια και το Κοινοβούλιο να απαιτήσει από το σύνολο των συναρμόδιων αρχών ε, τοπικές αρχές, περιφερειακές αρχές, Ευρωπαϊκή Ένωση να τους πούμε ότι θα πρέπει να κάνουν κάτι για ένα από τα πιο πολύτυπα πράγματα τα οποία έχουμε, όχι Ισπανία, Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα, τα, τα ποτάμια, αυτά τα ποτάμια, αυτούς τους κόλπους, τα, τα, τα εκεί πέρα, ε, τα γαλλικιανά τα οποία είναι πάρα πολύ πλούσια πλευράς ζωή, από πλευράς ε, ε, πανίδα χλωρίδα και επομένω πρόκειται για ένα μπλούτο, μια κληρονομιά. Και αυτό αφορά και τα μαλάκια, τα, τα θαλασσινά που ζουν εκεί πέρα. Επομένω θα πρέπει να υπάρχει μια ανταπόκριση στο, στο πρόβλημα αυτό. Και εκτός από τον φυσικό πλούτο, εκτός από τα οικονομικά, είναι και θέμα υγείας του κόσμου. Τέλος πάντων, κατάφερε η αποστολή να ανταποκριθεί σε αυτούς τους αγανακτισμένους και επίσης ε, είπαν οι αγνατισμένοι δεν θέλουμε να, να, να, έρθουν εδώ και να ανέβουν στα σκάφη μας οι αρχές γιατί νιώθουμε τέτοια αγανάκτηση. Εμείς τους δικαιώσαμε και τελικά σε συνεννόηση με τις αρχές μπορέσαμε να διαμεσολαβήσουμε κατά κάποιο τρόπο και καταφέραμε όλες οι βάσιμες ε, αναφορές, αυτές που κρεμούσαν τόσα χρόνια, να ε, πάνε προς την δικαίωσή τους, τη διεκπαιρέωσή τους. Επίσης θα πρέπει εκεί στα ποτάμια να γίνεται ολοκληρωμένη δουλειά. Δεν ωφελεί να καθίσουν τη μια πλευρά ή τη μια όχθη και όχι την απέναντι. Αυτό δεν είναι λύση του προβλήματο. Θα πρέπει όμω να είναι δύναμη, ε, λύση να δίνεται σφαιρική, συνολική. Και, και ε, είπα, είπαμε ότι αλλού είναι μεγάλο το πρόβλημα, αλλού μικρότερο. Α πούμε, στο Βίγκο υπάρχει ένα πρόβλημα, γι' αυτό γίνεται εκεί ζήμωση, προβληματισμό ε, για το αν θα κάνουν μικρές ή μεγάλες ε, εγκαταστάσεις για καθαρισμό του νερού, αν θα γίνουν σε δίκτυο τέλος πάντων αυτές οι εγκαταστάσεις. Ε, βρέχει πολύ στη Γαλλικία και θα πρέπει να δούμε κατά πόσον όλη αυτή η βροχή θα μπλεχτεί και θα εμποδίσει το έργο της του καθαρισμού των νερού. Στο Φερόλ, στο Φερόλ όντως η κατάσταση εκεί είναι η κατάσταση συναγερμού έχει χτυπήσει το καμπανάκι του Σαγερμού γιατί έχουμε μεγάλη υποβάθμιση εκεί του περιβάλλοντος. Και εκεί έχουμε την εγκατάσταση στην Ρεγανόσα. Δεν ξέρω γιατί. Κάποιος και κάποιο συμφέρον. Το κάτσανε και φτιάξανε την εγκατάσταση στο χειρότερο μέρος. Και γι' αυτό και φτιάξαν αυτές τις εγκαταστάσεις σε ένα μέρος που δεν πληρείται καμία προϋπόθεση ασφαλείας. Εκεί που χτίσαν το, τις εγκαταστάσεις, εκεί που είναι τα σπίτια τους, εκεί που έχει... Και αυτά τα μεγάφωνα, οι ντουντούκες εκεί για, κατάσταση ανάγκης. Ε, είναι, είναι, εντυπωσιακό το πώς το κάνανε έτσι. Ε, ας κάτσουμε να το σκεφτούμε λοιπόν σοβαρά. Και να πούμε σε κάποια έκθεση την γνώμη μας στον Μπούργο τώρα. Εκεί θα πρέπει όντω να, να, να γίνει μια έρευνα και εκεί θα πρέπει να αποφανθεί κάποιο και να δούμε πώ είναι δυνατόν η κατάσταση να βελτιωθεί, να λυθεί το πρόβλημα. Εν κατακλείδη. Πολύ σημαντική ήταν αυτή η αποστολή. Και για τη Γαλλικία και για την Ισπανία και για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα ολοκληρωμένα συστήματα τα συστήματα αποτελούν πλούτο, οικολογική κληρονομιά. Άρα κάτι το πολύ σημαντικό εγκατακλείδη. Όταν οι αρχές δεν δίνουν προτεραιότητα σε αυτού του είδους το, το, το, τις δημόσιες καταστάσεις, αυτό δεν είναι τυχαίο. Οι αρχές βάζουν άλλες προτεραιότητες και αυτό είναι λάθος. Πολύ μεγάλο λάθος. Είμαστε πολύ πίσω σε περιβαλλοντική νομοθεσία σε σχέση με άλλα κρατημέλη. Αλλά όταν και αυτά τα, λίγα νομοθετήματα που έχουμε δεν τα τηρούμε, τότε ε, το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Άρα, θα πρέπει να κάτσουμε να φτιάξουμε μια έκθεση. Ενδελεχή. Να είναι χρήσιμη και στον κόσμο και στις αρχές και να αρχίσουν επιτέλου οι αρχές, να βάλουν ένα χρονοδιάγραμμα για την επίλυση των προβλημάτων. Κύριε Μέγερ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Μπέρμαν, για του φιλελευθέρου έχετε δει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο, κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να τοποθετηθώ σε ορισμένα θέματα. Κατά την άποψή μου, η ε, επίσκεψη ήταν πολύ επιτυχημένη για διάφορους λόγους. Καταρχήν πρέπει να έχουμε κατά νου ότι το πρώτο που μας ενδιέφερε ήταν οι αναφέροντες με το αίτημά τους που ήταν ε, να λάβουμε υπόψη μας ε, αυτά τα προβλήματα. Εγώ έρχομαι από ορεινή περιοχή, από την Αυστρία. Έχω δει τη θάλασσα, αλλά ποτέ στη ζωή μου δεν έχω δει μαύρη θάλασσα. Αυτό που είδαμε βγαίνοντα από το λεωφορείο ήταν μια μαύρη θάλασσα. Πιάσαμε τη μύτη μα και όλοι λέγανε φρίκι, ούτε που θα ήθελα να ζω εδώ. Νομίζω λοιπόν ότι οι αναφέροντε πολύ σωστά μας επισήμαναν τι ακριβώ συμβαίνει. Επίση, ε, κατέστη σαφέ ε, ότι ήταν πολύ σημαντικό το ότι εμεί ω Επιτροπή Αναφορών ε, ασχολούμεθα με τα προβλήματα τη φύση, Όταν οι εκπρόσωποι των αρχών Λοιπόν μας λένε ότι είναι σε επικοινωνία με τους αναφέροντες. Μα τι επικοινωνία είναι αυτή όταν ένας εκπρόσωπος ε, θεσμικός λέει μπροστά στον αναφέροντα ότι αυτά που λέτε δεν ισχύουν. Και εμείς ε, τα είδαμε μόνοι μας. Είχαμε πετάξει τη θάλασσα, πολυθρόνες, ε, τηλεοράσεις, παλούκια, κομμάτια από σίδερο. Μα και εγώ τι να σκεφτώ, ότι είμαι τυφλή ή ότι βλέπω εφιάλτη. Νομίζω λοιπόν ότι το πρόβλημα που αφορά τις ε, σχέσεις ε, αρχών και αναφερόντων, προσπάθησα αυτό να το καταστήσω σαφές, το πρόβλημα είναι το εξή. Είναι θέμα επικοινωνία. Πώ επικοινωνούν αυτοί. Δηλαδή, όταν οι αρχέ λένε ότι επικοινωνούν με του αναφέροντε, οι αναφέροντε ε, παραπονιούνται ότι δεν του ε, λαμβάνουν υπόψη του. Εγώ πιστεύω του αναφέροντε. Προφανώ θα πρέπει οι αρχέ να μιλάνε με μία γλώσσα που να είναι κατανοητή από τον πολίτη. Αν βέβαια επιθυμούμε να βρούμε κάποια λύση. Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Ε, αναφέρθηκε επανειλημμένα και στην Ισπανία γιατί οι αναφέροντες ε, ε, δεν ε, κάλεσαν την τελευταία μέρα πάνω στο σκάφος και τους εκπροσώπους των αρχών. Ξέρετε γιατί δεν χώραγαν. Γιατί κάθε σκάφος μπορεί να δεχτεί μόνο ορισμένους επιβάτες. 11 ήταν ας πούμε και ένας. Ένας είναι ο καπετάνιος. δεν μπορεί αφού είναι 11 και ένας να μπει και 12 για λόγους ασφάλειας. Και αν το έκανε αυτό ο καπετάνιος, θα είχανε την άδειά του. Και δεν το ήθελε. Και σας το λέω, γιατί και εγώ έχω άδεια καπετάνιου και ξέρω πόσο αυστηρές είναι οι διατάξεις σχετικά με το πώς οι επιβάτες επιτρέπεται να ανέβουν σε ένα σκάφος. Κατά τα άλλα, να πω, το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα και το γεγονός ότι το συζητάμε εδώ, αυτό και μόνο είναι πολύ λυπηρό. Και δεν θέλω να πω τίποτα άλλο επ' αυτού. Ε, θέλω να δείξω και ένα άλλο θέμα. Τα διαρθρωτικά κονδύλια. Νομίζω όλοι μας ε, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι εδώ πρόκειται για χρήματα του Ευρωπαίου φορολογούμενου. Είναι χρήματα τα οποία σπαταλώνται και αυτό είναι απαράδεκτο. Εμείς ε, περιμένουμε από όλες τις αρχές, είτε είναι αυστριακές, γαλλικές, γερμανικές, δεν ξέρω εγώ ποιες, τέλος πάντων όλες να σκεφτούν ε, το πού θα ε, ανεγερθεί ε, μια τέτοια κατάσταση. Θα είναι αποτελεσματική, θα είναι φιλική προς τον πολίτη και αφού γίνουν οι σωστές σκέψεις, όχι μόνο θα προστατευτεί το περιβάλλον, γιατί είδαμε στο τέλος ότι είναι δυνατόν να, βελτιωθούν, ε, να βελτιωθεί το επίπεδο ε, των υδάτων, ε, να προσφερθούν θέσεις απασχόλησης και νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό μπορεί κανείς να προστατεύσει και το περιβάλλον, να αποφύγει όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στην Ευρώπη και σε άλλα μέρη. Κατόπιν τούτου νομίζω ότι Πρέπει να τα σκεφτούμε όλα αυτά. Ήταν επιγόντως απαραίτητο να επισκεφτούμε αυτή την περιοχή. Νομίζω δείξαμε ποιος μας ενδιαφέρει περισσότερο από όλους. Μα ο πολίτης. Και ξέρετε, αυτό δεν είναι μόνο ισπανικό πρόβλημα, το πρόβλημα του περιβάλλοντος αφορά όλους. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ και νομίζω ότι θα συντάξουμε μια πολύ καλή έκθεση. Πολύ καλά κύριε Μπέρμαν. Έχει ζητήσει τώρα λόγο ο κύριος Μιγιάν, ο κύριος ε, Μπουλό και παρακαλώ. παρακαλώ. Σύντομα. Ε, κάποιος άλλος επίσης ε, θα ήθελε να το Όχι, κύριε Μιγιάν. Όχι, εντάξει, εντάξει, μου, μου αρκούν τα δύο λεπτά. Μίλησα με τους ε, αναφέροντες. Μάρτυρες, η γραμματεία και ο πρόεδρος της αποστολής. και είπαμε ότι θα μπορούσε να, έρθει 11 να μας δείξει να έρθει ένας. Και είπαν δύο φορές, δύο φορές ήταν σε επαφή με αυτούς και από την Ένωση των Τσαράδων και από το, τη φορέα του, του, για το ποτάμι. Τέλος πάντων, το θέμα δεν ήταν να θα μπουν στο, στο σκάφος 11, 12 και 13. Αυτό που μου είπαν ήταν ότι δεν θέλανε, δεν θέλανε να έρθουν ε, από τις αρχές κάποιοι πάνω στο σκάφος. Τα ξέρει η γραμματεία, τα ξέρει ο πρόεδρος της, ε, της αποστολή μας. Έγινε, έγινε επίσημη επαφή. Και όταν μου λέγανε ότι δεν θέλουν, τότε και εγώ προσπάθησα και, προσωπικά. Ο ίδιος εγώ, όχι μέσω του Πρόεδρου. Ε, κοίτα και, και, και τον έναν και τον άλλον χωριστά. Μου απάντησαν όμως αρνητικά. Και είπανε ότι εάν ανέβουν οι αρχές στο καράβι, θα, θα, θα υπάρξει εκνευρισμός, θα, θα, θα υπάρχει εντεταμένο κλίμα. Και είπαμε ότι ε, καταλήξαμε ε, να το δούμε κάπως μονομερός, να δούμε μόνο εκεί κάτι, κάτι καλύβες, όπως λέμε για το... Ε, είχε κάτι, κάτι εξαθλειωμένους λαθρομετανάστες, κάτι, τη μαύρη τρύπα της περιοχής είδαμε. Επομένως, ξαναλέω, αυτό το πρόβλημα δεν ήταν επειδή έλειπε ο χώρος. Έλειπε γιατί ήταν τα πράγματα τα νεύρα, ήταν τεντωμένα Πάρα πολύ γρήγορα θέλω να σα πω, λέει ο πρόεδρο. να σα πω ότι στι 12.30 πρέπει να κλείσουμε. Στι 12.30 έχουμε μόνο μια μισή ώρα ακόμα. Μόνο μια μισή ώρα και έχουμε άλλε τρει, τρει, τέσσερι αναφορές. Ε, πάντων, νομίζω ότι υπάρχει ο χρόνο ούτω ώστε να μπορέσουν οι συνάδελφοι να έχουν το χρόνο που χρειάζονται. Κύριε Μπουλού Και μετά κύριε Μιράντα. Μάλιστα κύριε Πρόεδρε. Ναι, σας επιβεβαιώνω ότι και εγώ διαπραγματεύτηκα αυτό το σημείο της τελευταίας μας, του τελευταίου μας ταξιδιού. Οι αναφέροντες μου εξήγησαν ότι προτιμούσαν να τα πούν μεταξύ τους και μετά να μας παρουσιάσουν συλλογικά τα αιτήματά τους. Τους είπα ότι οι αρχές την προηγούμενη μέρα με το πλοίο μας είπαν ότι ε, ότι λέγω θα ήθελα να γίνουν αλλιώ τα πράγματα, αλλά τέλο πάντων δεν είναι σημαντικό πρόβλημα. Ελπίζω να μην χρειαστεί ολόκληρη ώρα να το συζητήσουμε. Κανείς δεν μας εμπόδισε να συζητήσουμε με τις τοπικές αρχές, άρα δεν πρόκειται για σοβαρό πρόβλημα. Ζήτησα όμως το λόγο για να πω και ζητώ συγγνώμη από τη γραμματεία που ξέχασα να το κάνω για την οργάνωση της επίσκεψης με όλα, με όλα, με τους διερμηνείς, διερμηνέτριες, τα τραπέζια, τα πλοία κτλ. Όπως είπαμε και πριν, στον τύπο αναφέρθηκαν όλα αυτά πολύ θετικά, εκτός από έναν τίτλο που έλεγε η Ευρώπη χρειάστηκε 15 χρόνια για να επισκεφθεί τη Γαλλική. Εκτός από αυτόν τον τίτλο, αν και το περιεχόμενο ήταν και αυτό θετικό, το σύνολο είχε θετική ανταπόκουρηση και έλεγε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έρχεται και ακούει τους αναφέροντες και τις αναφέρουσες. Και επειδή το 13 είναι το έτος Ευρωπαϊκής Ιθαγενείας, είναι πολύ καλό αυτό. Εχθές έγινε ο ακρόαση για την Ιθαγένεια και κατά τις συζητήσεις κάποιος εξέφρασε τη λύπη του γιατί λέει δεν υπήρχαν αρκετά μέτρα πρόληψης. Και στη Γαλλικία ισχύει αυτό, γιατί είδαμε κατά την επίσκεψη αυτή ότι τα οι που δεν ήταν πρόληψη ήταν παρόλα, είχαν παρόλα αυτά θετική επίπτωση και οδήγησαν στη λήψη μέτρων. Άρα και τα τιμωρητικά μέτρα είναι αποτελεσματικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει διαρθρωτική ποσά από τα διαρθρωτικών ταμείων και στη Γαλλική όχι μόνο για το περιβάλλον, αλλά για τη συνολική οικονομική ανάπτυξη για την αλληλεία, τον τουρισμό, την βιώσιμη ανάπτυξη, την υγεία, για όλα αυτά, για όλα αυτά διαθέτει πως ακόμη κι αν σε ορισμένες περιπτώσεις οι τοπικές αρχές σέβονται μόνο εν μέρη τις οδηγίες. Αν μπορούμε λοιπόν να κάνουμε κάτι ώστε η αναθέρμανση της αλληλείας εκεί να μπορέσει να βελτιωθεί, να γίνει, τόσο το καλύτερο. Λοιπόν, για... η επίσκεψη έπρεπε να γίνει με πολύ μεγάλη ταχύτητα γιατί η... απαερημένουμε ακόμη τις απαντήσεις των ερωτημάτων που είχαμε θέσει στις τοπικές και περιφερειακές αρχές και που τις χρειαζόμαστε για να κάνουμε την έκθεσή μας. Τέλος, σεβαστήκαμε την, τα Πήγαμε να προσκυνήσουμε τον Άγιο Ιάκωβο της Κομποστέλης και ελπίζω η τελική έκθεση να εγκριθεί λοιπόν ομόφωνα και να ικανοποιήσει και την Γαλλικία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και συμφωνώ 100% με αυτά που είπε ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας μας ότι δεν θα πρέπει να κολλάμε στις λεπτομέρειες. Πρόκειται για έκθεση πολύ σημαντική, ε, αφορούσε πάρα πολύ κόσμο και είναι συμφέρον των αρχών να υπάρξει τελικά κάποιος διάλογος και οι λεπτομέρειες ποιος, πότε, γιατί ε, δεν μπορεί να ανέβει στο σκάφος είναι το, το, το δέντρο που είναι το δέντρο που βλέπουμε αντί να δούμε το δάσο. Τα, τα είπε ο πρόεδρο σωστά και πραγματικά έτσι ήταν τα πράγματα ε, και τελικά κάποιοι νιώθανε ε, άβολα γιατί είδαμε ότι οι αρχές που μπορούσαν να κάνουν αυτό το οποίο κάνανε όπως μας τα είπανε και, και ο σύμβουλος και, και η σύμβουλος τέλος πάντων όλοι αυτοί υποτίθεται ότι πρέπει να ξέρουν το πρόβλημα. και η περιοχή που αφορά το πρόβλημα είναι η περιοχή όπου κάποτε ε, μάζευαν όλα εκείνα τα θαλασσινά, τα, τα κοχύλια, τα, τα, τα μύδια, όλα τέλο πάντων τα, τα, τα, σχετικά, τα θαλασσινά. Και επομένως αυτός που ξέρει τον Μπουργκό, αυτός που ξέρει ε, για αυτό, αυτό τον κόλπο, ε, ξέρει ότι εκεί είναι κατεξοχήν η μόλυνση. Οπότε πριν κανεί ε, έχει άποψη πρέπει να πάει και να δει που τι γίνεται. Ευχαριστούμε κύριε Μιάννα, λέει ο Πρόεδρο. Οπότε ολοκληρώσαμε αυτό το θέμα και ε, θα ήθελα να σα πω ότι και, και εγώ έχω πάει εκεί πέρα και όπω είπατε ήταν όντω μικρό το σκάφο. Είχαμε του ε, διερμηνεί, είχαμε τη γραμματεία, ε, δεν χωράγανε κι άλλοι. Θα έπρεπε να λυθεί το πρόβλημα με άλλο σκάφο. Είχαμε κι άλλο Έχαμε διαλέξει ένα πιο μεγάλο τέλος πάντων. Πρόκειται για θέμα για το οποίο μιλήσαμε και τα είπαμε. Τώρα, πάμε στο σημείο υπαριθμών 9. Η γνωμοδότηση για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Για κάποια σχέδια δημόσια και ιδιωτικά και τις επιπτώσεις του στο περιβάλλον. Είναι εισηγητής ο κύριος Χουντής. Έχουμε κάποια πρώτη ανταλλαγή απόψεων τώρα και θα έχει το λόγο ο κύριος Χουντής. Έχετε τον ε, λόγο κύριε Χουντή. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. because he has arrived the president and we are in the no, number okay, nine okay. and can, we start. You can start. Μπορείτε αρχίστε κύριε Χουντή, μπορείτε αρχίστε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ωραία. Σας ευχαρίστησα και εσά και τον προηγούμενο πρόεδρο. Ε, ε, σας παρακαλώ απαντήστε μου στην εξής ερώτηση. Πόσο χρόνο διαθέτω. Πόσο χρόνο έχω γιατί η, η διαχείριση του χρόνου φαίνεται ότι είναι πρόβλημα. Ναι. Πόσο χρόνο ε, μου δίνετε για την παρουσίαση της γνωμοδότησης. Ε, I think five minutes, but if you something else, Ωραία. You can. Ναι, καθαρές κουβέντες. Λοιπόν, okay. ωραία, ωραία. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, είμαστε στη δεύτερη συζήτηση της γνωμοδότησης για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Πριν επαναλάβω ορισμένες από τις βασικές παρατηρήσεις που είχα καταθέσει κατά την πρώτη συζήτηση με αρκετές με, ε, με προσθήκες, θέλω να σας πω ότι από τη συζήτηση ε, από την πρώτη συζήτηση που είχαμε κάνει είχα διατυπώσει και ενισχύθηκε το αίτημα από όλους σχεδόν τους ομιλητές, από όλες σχεδόν τις ομάδες ότι θέλουμε περισσότερο χρόνο για να δουλέψουμε. Υλοποιώντας την εντολή λοιπόν της Επιτροπής συναντήθηκα με τον ε, εισηγητή από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, τον κύριο Ζανώνη. Εκεί κάναμε κουβέντα για όλα τα θέματα και για το σχετικό ε, αίτημα και με τη συνδρομή της ε, συνεργάτη μου της κυρίας Πανταζίδου που είναι δίπλα μου και του κυρίου David Lott, David από τη Γραμματεία με τη συνδρομή τους και τα επιχειρήματά τους τον πείσαμε τον εισηγητή και μας έδωσε ένα μήνα παράταση. Σας παρακαλώ λοιπόν προσέξτε όπως βλέπω έχει τροποποιηθεί λοιπόν το πρόγραμμα και είμαστε σύμφωνοι Δηλαδή θα ψηφίσουμε τέλη Ιουνίου και όχι τέλη Μαΐου όπως αρχικά έλεγε το χρονοδιάγραμμα. Για μένα παραμένει ένα ερώτημα, πρέπει να, με να συνοηθούμε με τη γραμματεία, πότε πρέπει να κατατεθεί το κείμενο για να μπορέσει να μεταφραστεί και να το πάρουν οι συνάδελφοι, πείτε μου την ημερομηνία στο τέλος. Μπαίνω λοιπόν στην ουσία, εφόσον διευκρινίσαμε αυτά τα θέματα, ε, θα τα εξαντλήσω τα πέντε λεπτά όσο γίνεται πιο γρήγορα. Νομίζω ότι για τη σημασία ε, που, έχει η τροποποίηση που γίνεται για την γνωμοδότηση, ε, η τροποποίηση που γίνεται για την οδηγία που αντιμετωπίζει τα ζητήματα περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχουμε συζητήσει και συζητήσαμε και αρκετές φορές. Προσθέτω, στο μεσοδιάστημα που συζητήσαμε η εμπειρία η ελληνική και ενδεχομένως και από άλλες χώρες μου επιβεβαιώνει ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμα τα θέματα. Και ακόμα Θέλω να σας πω ότι επειδή η πληροφόρηση ότι τροποποιείται η οδηγία και αφήνει περισσότερα περιθώρια για παραβιάσεις και εξαιρέσεις ήδη έχει διαχυθεί. Δηλαδή πριν εγκριθεί η οδηγία ήδη κινούνται ορισμένοι με βάση εξαιρέσεις, ορισμένες εκ των οποίων εγώ δεν συμφωνώ και θα το επαναλάβω. Επομένως είναι μια ζωντανή διαδικασία έτσι κι αλλιώς και σας εφιστώ για άλλη μια φορά την προσοχή αν μου επιτρέπετε αυτό. Τώρα, <clears throat> μπαίνω στις, βασικές, στις βασικότερες τροποποίησεις για να ξεκινήσει πάλι η συζήτησή μας. Το πρώτο, η πρώτη παρατήρηση είναι ότι είναι θετι... ορισμένα τα θετικά τα τονίζω, δεν τα χαρακτηρίζω πάντα. Είναι θετικό ότι τίθεται το θέμα της βιοποικιλότητας στο άρθρο 3 και στα παραρτήματα. Ε, θα καταθέσω τροπολογία για το σαφή ορισμό της βιοποικιλότητας με βάση τη συνθήκη για τη βιολογική ποικιλότητα. Δηλαδή τι σημαίνει ο όρος βιοποικιλότητα. Δεύτερο, ε, οι εξαιρέσεις όπως σας ανέφερα πριν, ως μια ζωντανή κατάσταση που διαχέεται ήδη στην πρακτική εφαρμογή, εφαρμογή ε, αποδυναμώνουν την οδηγία. Μένω και υπογραμμίζω ότι προτείνω να διαγραφεί από το άρθρο 1 η παράγραφος 4 σύμφωνα με την οποία η οδηγία δεν, η οδηγία δεν εφαρμόζεται για έργα που εγκρίνονται με ειδική εθνική νομοθετική πράξη. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο, απλώς θυμίζω την παρατήρησή μου ότι αρκετές χώρες, ιδιαίτερα αυτές που βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, μέσα στους αναπτυξιακούς στόχους περιλαμβάνουν fast track διαδικασίες που παρακάμπτουν τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και την προστασία, στο όνομα να κάνουμε γρήγορα ανάπτυξη. Τρίτο, ε, νομίζω ε, μάλλον είμαι αντίθετο στην πρόταση ότι τα πληροφοριακά στοιχεία πρέπει να τα δίδει ο κύριο του έργου, Αυτό που θα δίνει, θα αναλαμβάνει το έργο και θα δίνει διάφορες πληροφορίες και τα λοιπά και τι επιπτώσει ενδεχομένω έχει στο περιβάλλον και όχι, και εκείνη η διαφωνία μου, να μην παρουσιάζονται και εναλλακτικέ λύσει. Διότι κατά αυτή την έννοια θα λέει είναι αυτό, θα έχουμε αυτέ τι επιπτώσει, θα τα διορθώσουμε. Ενώ δεν θα έχουμε μπροστά μα εναλλακτικέ προτάσει που θα μπορούσαμε να τι είχαμε αποφύγει. Και βεβαίως εδώ είναι και ο ρόλος και τη συμμετοχής των πολιτών, του κοινού. Ε, επίσης, θεωρώ ότι αυτό το ζήτημα της συμμετοχής του κοινού σε όλες αυτές τις διαβουλεύσεις, σε, όλες, σε όλα τα βήματα για να μην αναφερθώ αναλυτικά, από τη συζήτηση οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής, scoping, έτσι το βρήκα και εγώ αυτή την ορολογία ίσως για να γίνει κατανοητό, δηλαδή διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές, θα πρέπει να εξασφαλιστεί και από αυτή την φάση της διαδικασίας η συμμετοχή του κοινού. Ε, για την ενίσχυση αυτής της διαδικασίας ε, ε, νομίζω ότι, και θα το τονίσω, η οδηγία πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνη με τη σύμβαση του Άορχους που περιλαμβάνει την πρόσβαση σε πληροφορίες με τη συμμετοχή του κοινού. Ένα άλλο σημαντικό σημείο, δεν θα σας κουράσω πολύ, είναι οι επανειλημμένες συζητήσεις για τις μελέτες ε, περιβάλλοντος, επιπτώσεις ε, στο, περιβάλλον, οι οποίες στερούνται, μάλλον έχουν γίνει κατά κανόνα αναξιόπιστες. Και έχουν γίνει κατά κανόνα αναξιόπιστες διότι τη σύνταξή τους ανατίθεται στον κύριο του έργου. Η πρόταση είναι να μην την έχει αυτός, να, έχουν, να την έχουν ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες και μάλιστα πάω και λίγο παρακάτω, αν αποδεδειγμένα η μελέτη που κάνουν, γιατί έχει αποδειχθεί, αυτοί οι εμπειρογνώμενες όσο αφορά τις επιπτώσεις είναι λαθεμένες, να επιβάλλονται και κυρώσει και σε αυτού του κυρίω, διότι πολλέ φορέ, τι περισσότερε φορέ, τα προβλήματα ξεκινάνε από εσφαλμένε ή με ελλειπή στοιχεία ή με ελλείψει, όπω χαρακτηρίζεται μετά κατά την κοινοτική νομοθεσία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ε, τελειώνω με, το, με δύο σημεία ακόμα. Είναι θετικό ότι προβλέπεται να υπάρχει ένας μηχανισμός παρακολούθησης των επιπτώσεων κατά την εφαρμογή του έργου ε, όμως το θέμα είναι αυτό, ε, αν αυτός ο μηχανισμός θα δίνει τη δυνατότητα στην αρμόδια αρχή να επεμβαίνει διορθωτικά και να σταματάει πιθανόν εκτελούμενο έργο αν έχει τέτοιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τέλος, αναφέρομαι στο θέμα της εξόρυξης σχιστολιθικού φυσικού αερίου και σχιστολιθικού πετρελαίου, ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει και για άλλους λόγους. Προτείνω ε, επειδή έχει επικίνδυνες επιπτώσεις στο νερό, στη βιοπικιλότητα κτλ. Προτείνω ε, να συμπεριληφθούν αυτές οι επιπτώσεις στο παράρτημα 1 της οδηγίας ώστε να αξιολογούνται σωστά και να λαμβάνονται υπόψη. Αυτές είναι οι βασικότερες παρατηρήσεις. Ε, επαναλαμβάνω, περιμένω και από τη γραμματεία πότε ε, θα πρέπει να κατατηθεί το κείμενο για μετάφραση και περιμένω ο, με ενδιαφέρον τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις των συναδέλφων. Ευχαριστώ. Εξάντησα το πεντάλεπτο, αλλά δεν θα το κάνω στη δευτερολογία, αν χρειαστεί, να το συντομεύσω. Ευχαριστώ. Thank you to you. You were perfect. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια χαρά τα είπατε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την Επιτροπή, τον κύριο Στέφανο Αμπατζή. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος ε, να τοποθετηθώ ε, άμεσα στα θέματα που έθιξε ο κύριος Χουντής. Και εγώ επίσης ε, συμφωνώ ότι η σημασία αυτής της οδηγίας δεν χρειάζεται πλέον να προβληθεί και περνάω στα διάφορα θέματα επί της ουσίας. Όσον αφορά λοιπόν τις δυνατότητες εξαίρεσης ή παραβίασης, η Κομισιόν δεν συμφωνεί με αυτή την παρατήρηση. Πιστεύει ότι θα πρέπει να ε, ε, ενισχύσουμε περισσότερο την ποιότητα της οδηγίας και με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί και το επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας. Και όσον αφορά τις δύο εξαιρέσεις που έχει κατά ο κύριος ε, Χουντής, άρθρο 1, παράγραφος 3, αυτό που λέει η Κομισιόν είναι ότι οι εξαιρέσεις πρέπει να είναι πιο αυστηρές από ό,τι είναι σήμερα. Αν δείτε λοιπόν τη σχετική τροπολογία, έχουμε καταθέσει εμείς μια τροπολογία που λέει ότι ε, είναι δυνατόν να υπάρχουν εξαιρέσεις μόνο εφόσον ο στόχος ε, είναι η εθνική άμυνα ε, ή κάποια άλλη μορφή προστασία. Αυτό το αποκλειστικά και μόνο δεν υπάρχει, αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών. Άρα δηλαδή λέμε να περιοριστεί αυτό. Όσον αφορά την διαγραφή του 1-4, εδώ δεν πρόκειται κατ' ουσίαν για εξαίρεση. Στην παράγραφο 1, σημείο 4, εκεί αναφέρεται ότι όταν το Κοινοβούλιο ενός κράτους μέλους εγκρίνει ένα πρόγραμμα, τότε οι στόχοι της οδηγίας πρέπει να γίνονται σεβαστοί και για να υπάρχει ασφάλεια ότι τα κράτη-μέλη δεν κάνουν κατάχρηση, εμείς ε, λέμε ότι υπάρχει υποχρέωση λογοδοσίας από πλευράς κατων μελών που καταφεύγουν σε αυτή τη διάταξη. Άρα δηλαδή το θέμα δεν είναι εξαιρέσεις ή παραβιάσεις, το θέμα είναι πού τις εντάσσουμε όλες αυτές, μέσα σε ποιο πλαίσιο. Όσον αφορά τώρα τη βιοπικιλότητα, πράγματι και εγώ συμφωνώ ότι είναι απαραίτητο να οριστεί η βιοπικιλότητα. Αλλά εμείς στην πρόταση της Επιτροπής ε, προσπαθήσαμε να μην ορίσουμε εμείς θέματα για τα οποία υπάρχει ήδη διεθνής ορισμός. Ας πούμε, στο εδάφιο 7 κάνουμε αναφορά στο ε, στη σχετική σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, όπου εκεί υπάρχει ορισμός του όρου βιοπικιλότητα. Άρα δηλαδή αν δεν υπάρχει δικό μα ορισμό, το εδάφιο υπερτμών 7 ήδη καλύπτει το θέμα αυτό και σα το επισημαίνω. Όσον αφορά τώρα τις πληροφορίε που πρέπει να ε, υποβάλει ο κύριος του έργου ε, και σχετικά με τις αναλλακτικέ λύσεις, αυτό είναι δική μα ε, σημαντική πρόταση και προτείνουμε ο κύριος του έργου όταν προετοιμάζει την έκθεση δεν προτείνει πλέον εκείνος τις εναλλακτικέ λύσεις, αλλά θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτική αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων σε σχέση με ένα έργο. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα καθοριστική σημασία θέματα, όπου προσπαθήσαμε να εξαλείψουμε τις δυναμίες της οδηγίας και αυτό το θέμα των εναλλακτικών λύσεων υπάρχει ήδη στην αρχική φάση και η Κομισιόν προτείνει η αρμόδια αρχή ο κύριος του έργου και επίσης και οι υπερβαλλοντικές αρχές στην αρχή της διαδικασίας να ορίζουν μόνοι τους ποιε είναι οι εναλλακτικέ λύσεις του project. Και επίσης ε, στο παράρτημα 4 αναφέρουμε ότι είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί και η μηδενική λύση, αυτό που λέμε baseline σενάριο, όπως ε, επίσης ε, και τις βέλτιστες εναλλακτικές λύσεις για ένα έργο. Πιστεύω λοιπόν ότι το θέμα των εναλλακτικών ε, λύσεων εξετάζεται ικανοποιητικά από την Κομισιόν. Όσον αφορά τώρα αυτό το περίφημο scoping και την ανάγκη ε, συμμετοχής. Το scoping γίνεται τώρα υποχρεωτικό και ενημερώνεται το κοινό, ενημερώνονται οι πολίτες αλλά δεν προβλέπεται, προβλέπονται υποχρεωτικές διαβουλεύσεις με τους πολίτες σε αυτή τη φάση. Οι πληροφορίες που δίδονται στο πλαίσιο του scoping διοχετεύονται στους πολίτες, αλλά δεν προβλέπονται διαβουλεύσεις. Ε, κατά τη δική μας την άποψη, αυτό είναι ένα θέμα διοικητικού αχθούς και φόρτου, λοιπόν, γι' αυτό δεν περιλαμβάνεται στην πρόταση της Κομισιόν. Όσον αφορά την πρόταση της EIA, Νομίζω ότι εδώ συμφωνούμε με αυτά που προτείνει ο εισηγητής, ε, παράγραφος 5, C, της πρότασης και μία από τις αναλλακτικές λύσεις είναι να έχουμε διαπιστευμένους και πιστοποιημένους εμπειρογνώμονες που θα καταρτίζουν τις εκθέσεις της EIA και υπάρχει και άλλη μια πρόταση πιο κάτω που λέει ότι εναπόκειται στα κράτη-μέλη να ορίσουν τα προσόντα αυτών των εμπειρογνωμόνων, πώς θα ε, καταχωρίζονται αυτοί οι εμπειρογνώμονες και εάν θα προβλέπονται κυρώσεις για αυτούς τους εμπειρογνώμους. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ συμφωνούμε ε, με τον εισηγητή και όσον αφορά τελικά το σχιστόλιτο Πρόκειται για μια οδηγία με 200 κατηγορίες. Ε, η τροποποίηση του παραρτήματος 1 δεν είναι πρόταση της Επιτροπής. Από την άλλη βέβαια, αν διαβάσετε λιγάκι τα κριτήρια που έχουμε στο παράρτημα υπαριθμών 3, είναι πολύ σημαντικά για τα προγράμματα εξόριξης ε, σχιστολίτου. Αναφερόμεθα σε επικίνδυνες ουσίες, στον κίνδυνο ε, μόλυνσης των υδάτων. Αυτά λοιπόν τα κριτήρια είναι καθοριστική σημασία για να ε, ξεκαθαρίζεται τι θα γίνεται με το σχιστόλιτο. Στο παράρτημα 4, εκεί υπάρχουν συγκεκριμένε ε, τροπολογίε που είναι πολύ σημαντικέ για το σχιστόλιτο. Πράγματι, λοιπόν, η πρόταση επιτροπή δεν περιλαμβάνει τίποτα συγκεκριμένο για το σχιστόλιτο, αλλά υπάρχουν άλλα θέματα που είναι συναφή. Για το σχιστόλιτο θέλω να σα πω ότι φέτο η Επιτροπή θα καταθέσει μια συγκεκριμένη πρόταση, ειδικά για το σχιστόλιτο. Γι' αυτό, λοιπόν, δεν υπάρχει παράρτημα, δεν υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση για το παράρτημα 1 και το παράρτημα 2. Ευχαριστώ. Oh, κυρία εν συντομία, μια που δεν έχουμε στα χέρια μας την έκθεση, να τονίσουμε ότι θεωρούμε ότι το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν θεωρούμε ότι υπάρχουσα οδηγία είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι. Οπότε ωραία να μα τα λέει αυτά η Κομισιόν, αλλά εγώ ασφαλή δεν αισθανόμαι. Μα λέτε για την παλιά ρύθμιση. Να το δούμε και στο επόμενο σημείο, στην επόμενη αναφορά όμω είναι σαφέ ότι από την συμφωνία, τη σύμβαση του Άρχου δεν έχετε καταλάβει τίποτα και μα λέτε για την παλιά. Εγώ οπότε αισθάνομαι ανασφαλή, φοβισμένη. Λέμε για αναθεώρηση της τροποποίησης οδηγία, ε, γιατί ο κόσμο ανησυχεί πάρα πολύ Πολύ περισσότερο από εσά. Εμεί εδώ τον κόσμο εκπροσωπούμε. Είμαστε μια επιτροπή που είναι κοντά στον κόσμο. Και η συμφωνία του Άρχους είναι πολύ πιο φιλική, α το πούμε, πολύ πιο κοντά στον κόσμο. Και το ξέρει αυτό ο κόσμος, ο πολίτης και ανησυχούμε πάρα πολύ για το μέλλον αυτή τη οδηγία. Και γι' αυτό ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να έχουμε κάποιο είδου αυστηρότερη, κάποιο είδου μεγαλύτερη ενάργεια τέλο πάντων από εσά. Η Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε. Κύριε Μποστινάρο. Madam Chair, I'm not completely happy and satisfied with the answers provided by the Commission. Because δεν μας δεκαπλώνει πόσο μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. For my very distinguished colleague Margaret Auken, if Aarhus Convention would be... Καλά είπε κύριε Auken. Εντάξει, άμα ήταν όλα τέλεια της του Άρχους δεν θα είχαμε σήμερα προβλήματα. Όμως έχουμε ένα νομικό πλαίσιο. Αυτό το οποίο υπάρχει ε, θα πρέπει να μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Αλλά αν ήταν έτσι πάλι δεν θα είχαμε τόσες και τόσες αναφορές οι οποίες αφορούν την παραβίαση της οδηγίας για, την, για τις μελέτες των περιβαλλοντικών επιπλώσεων. Επομένως είναι σαφές ότι κάτι πάει στραβά και όχι μόνο στη Δανία. Κάτι πάει στραβά με αυτή την οδηγία. Και άρα θα πρέπει να το διορθώσουμε. Ούτε πήραμε καμία απάντηση για σημεία πολύ σημαντικά πρώτα-πρώτα. Να ξεκάθαρο ορισμό. Πότε χρειάζεται στρατηγική μελέτη επιπτώσεων. Σχώς. Α, για αυτή τη σαλαμοποίηση. Τη γνωστή. Πότε χρειάζεται. Πρόκειται για επιπτώσεις πολύ σημαντικές. Μεγάλης κλίμακας. που πολλές φορές ε, πρόκειται για διατάξεις που τις παρακάμπτουν οι επενδυτές. Πώς θα εξασφαλίσουμε αυτή η μελέτη να είναι ουδέτερη, αμερόληπτη, αντικειμενική. Γιατί μιλάμε τώρα για μεγάλα προγράμματα, μεγάλα έργα τα οποία υποτίθεται ότι έχουν πολύ σοβαρές επιπτώσεις. Οπότε Πάντοτε τα καταφέρνει ο επενδυτής να παρακάμψει την ομοθεσία. Επομένως χρειάζεται να υπάρχει ένας σαφής ορισμός. Αν δεν υπάρχει σαφής ορισμός, πάντα ο επενδυτής θα βρίσκει κάποια εταιρεία, ούτω ώστε να τα καταφέρει με τον πιο φτηνό τρόπο. Να βρει τον αδύνατο κρίκο. ή πολλέ φορέ έχουμε τη μελέτη που λέει ότι όλα γίνανε καλά και στρογγυλά, αλλά το πρόβλημα υπάρχει. Άλλη τώρα... Άλλη μια ιδέα μου είναι για αυτή την, ε, τη, διασυνοριακή διάσταση, γιατί ξέρουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει κάποιο έργο το οποίο αναπτύσσεται, γίνεται στη Ρουμανία, αλλά μπορεί να έχει επιπτώσεις στην Ουγγαρία ή στη Βουλγαρία ή το αντίστροφο ας πούμε, και μεταξύ Τσεχίας και Γερμανίας. Αυτό πώς το αντιμετωπίζετε, αυτή την διασυνοριακή διάσταση του προβλήματος, γιατί πολλές φορές η εταιρεία η οποία κάνει τη μελέτη των επιπτώσεων θα εξετάσει μόνο, μόνο, μόνο, μόνο το, το, ένα κράτος. Δεν θα κοιτάξει τι είναι από μια μεριά των συνόρων. Να σας δώσω και ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Κάτι που, που το έλεγε το λέει και αναφορά. Θυμάστε αυτή την εταιρεία. Η Ουγγρική κυβέρνηση επισήμως είχε ζητήσει από την κυβέρνηση της Ρουμανίας να τους δοθούν όλες οι πληροφορίες ούτως ώστε να μπορέσουν και να υπολογίσουν την περιβαλλοντική επίπτωση. Σύμφωνα με την συνθήκη του Άρχους. Μιλάω για τη χώρα μου που η τότε κυβέρνηση αρνήθηκε να παράσχει την δέουσα ενημέρωση. Επομένως, και δεν έγινε και τίποτα. Πώς θα αποτρέψουμε τέτοιες καταστάσεις στο μέλλον, θα πρέπει να καλύψουμε και αυτή τη διάσταση. Το τι γίνεται με τη μεριά των συνόρων για τα μεγάλα έργα και προγράμματα. Τέλος. Πάρα πολύ ε, χαροποιεί αυτό το οποίο είπατε για το σχηματικό αέριο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ σωστό. Και επομένω ήρθε η ώρα να μπορέσουμε να έχουμε και μια οδηγία για το σχηματικό αέριο. Και επίση και εδώ εμπλέκεται η χώρα μου. Υπάρχουν εγκρίσεις και άδειες στην Νότια Ρουμανία για τέτοια εκμετάλλευση, αλλά είναι δυνατόν να υπάρχουν επιπτώσεις στα υπόγεια ύδατα, τα οποία υπόγεια ύδατα δυστυχώς ή ευτυχώς πάνε και πέρα από τα σύνορά μας. Πάνε στη Βουλγαρία. Και έτσι και εκεί ο τροφό ορίζοντα επηρεάζεται. Τι θα κάνουμε με το διασυνοριακό θέμα για να μην κυριαρχούν οι μεγαλοπενδυτές, οι πολυεθνείς, οι πολυεθνικές, συγγνώμη, εκείνοι οι οποίοι έχουν συνηθίσει να ασκούν πιέσεις. Τέλος πάντων είναι πάρα πολύ θετικά όλα αυτά τα οποία συζητούμε τώρα εδώ γιατί ήρθαν σε επαφή, μου, με σε επαφή μαζί μου η παραγωγή ε, ασχολούμενοι τόσο με τον κλάδο του σχεδιωτικού αερίου και του, του πετρελαίου και μου είπαν ότι θα πρέπει όλα αυτά να ληφθούν τώρα υπόψη. Γιατί αυτά είναι τα προβλήματα της Ένωσης, τα ουσιαστικά. Επομένως, αντιμετωπίστε τα αυτά. Αλλιώ δεν θα λύσουμε κανένα πρόβλημα. Ευχαριστούμε κύριε Μποστινάρου. Ναι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να κάνω μία, δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι η εξή. Η έκθεση αυτή είναι πολύ σημαντική για μας. Γιατί κατά την άποψή μου αυτό που είναι απολύτως απαραίτητο είναι να υπάρξει εναρμόνιση κατά την εκτέλεση στα κράτη-μέλη. Αυτό που είπε ο κύριο Μποστινάρου ε, και το έχω εγώ έτσι αρνητικά καταγράψει στο μυαλό μου, είναι ότι όταν έχουμε διασυνοριακά προγράμματα, περιβαλλοντικά προγράμματα, τότε μόνο καταλαβαίνει κανείς ε, πόσο διαφορετική είναι η εκτέλεση των διατάξεων και η εκτέλεση των έργων στα κράτη-μέλη. Άρα δηλαδή πρέπει να υπάρξει βελτίωση. Και σήμερα θα έχουμε άλλη μία αναφορά που αφορά το πρόβλημα ανάμεσα στην Τσεχία και τη Γερμανία και το ερώτημα που τίθεται είναι τι γίνεται όταν οι αρμόδιες αρχές καταλήγουν σε εκδιαμέτρου αντίθετες απόψεις. Μα δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό, αλλά δηλαδή κάτι δεν πάει καλά. Αυτό μιλάει από μόνο του. Ε, και νομίζω λοιπόν θα πρέπει ο εισηγητής ε, και οι σκιώδεις εισηγητές να ξανασυναντηθούν γιατί εδώ πρέπει να διατυπώσουμε βασικές πολιτικές θέσεις για να επιτύχουμε βελτίωση. Εγώ πιστεύω, ανεξάρτητα με το τι θα συμφωνήσουμε, θα πρέπει να υπάρχει εναρμόνιση. Δηλαδή, στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο να εφαρμόζονται οι ίδιες διαδικασίες, αλλά να ισχύουν επί του περιεχομένου και οι ίδιοι κανόνες πόσο μάλλον στα διασυνοριακά προγράμματα, γιατί ακριβώς σε αυτά ε, καθίστανται σαφείς οι ελλείψεις. Άρα δηλαδή εγώ προτείνω συγκεκριμένα να συναντηθούμε εισηγητής ε, και οι εισηγητές να την ξαναδούμε την έκθεση για να κάνουμε καλύτερες προτάσεις διατύπωσης. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ζήτησε κανείς άλλος να λάβει το λόγο. Νομίζω λοιπόν ότι ήταν ε, χρήσιμη αυτή η συζήτηση. Όλα αυτά που είπατε θα συμπεριληφθούν ε, στο σχέδιο εγγράφου ε, το οποίο θα συνταχθεί. Ο κ. Χουντή, ζητείτε το λόγο κύριε Χουντή, τον έχετε. Υποσχέθηκα ότι θα είμαι σύντομος και θα είμαι. Και η δεύτερη συζήτηση εδώ στην Επιτροπή μας μου επιβεβαίωσε πρώτον ότι η Επιτροπή μας αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα αυτής της οδηγίας και της τροποποίησης που επίκειται αντιλαμβάνεται ή τουλάχιστον η δική μου ερμηνεία είναι ότι μπροστά στη φάση της κρίσης μπορεί να γίνει ένα ιστορικό πισωγύρισμα στην κατά θετική περιβαλλοντική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργώντας αρνητικά συναισθήματα στους πολίτες που μέχρι τώρα περηφανεύονταν για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και εδώ υπάρχει η ανησυχία ότι πάμε πίσω. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Και το τρίτο, επιβεβαίωσαν την κατεύθυνση προς τα οποία πρέπει να κινηθούμε και να κινηθώ ως εισηγητής δίδοντας το, τις γραπτές προτάσεις για να μπορούμε να μιλάμε πιο συγκεκριμένα και να μπορούμε να κάνουμε την συζήτησή μας πιο ουσιαστικά. Προς το παρόν μοιάζει ένας διάλογος με την Επιτροπή και από τα σημεία που έθιξε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής ε, θα μπορούσα να πω ορισμένα ένα μόνο θέμα. Με ανησυχούν γενικώ οι εξαιρέσεις. Ε, εγώ αναφέρθηκα σε άλλη εξαίρεση και όχι σε αυτή που απάντησε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Δεν αναφέρομαι στην εξαίρεση του σημείου 3 του άρθρου του 1 σχετικά με ειδικέ συνθήκες πολιτικής προστασίας. Δεν αναφέρθηκα σήμερα σε αυτό. Πράγματι, εν πάση περιπτώσει, στην αρχική οδηγία δεν υπάρχει τέτοια διάταξη. Τίθεται εκεί. Να το βάλουμε όμως με πολύ πολύ αυστηρούς όρους, διότι στο όνομα ειδικών καταστάσεων, ειδική ανάγκης πολιτικής προστασίας μπορεί να γίνουν σημεία και τέρατα και μπορώ να σας πω παραδείγματα. Όμως, σήμερα αναφέρθηκα στην εξαίρεση που γίνεται για έργα που ρυθμίζονται ή για τα οποία υπάρχει ειδική εθνική νομοθετική πράξη. Και εδώ έγκυται οι μεγαλύτερες ανησυχίες μου. Διότι σε αυτή τη φάση έχω πολλά παραδείγματα που τα εθνικά κοινοβούλια νομοθετούν κατά παραβίαση εθνικών συνταγμάτων, κατά παραβίαση κοινοτικού δικαίου, προκειμένου να πετύχουν ορισμένους στόχους που τίθενται μέσα από τη δημοσιονομική εξυγίανση κτλ. Με ανησυχεί αυτή η διαδικασία την οποία τώρα θα επικαλεστούμε ως εξαίρεση για να περάσουμε πράγματα που δεν θα τα επιθυμούσε κανένας. Εκεί έγκυται η μεγαλύτερη μου ανησυχία και εκεί θα χρειαστεί να το συζητήσουμε πιο συγκεκριμένα. Σε κάθε περίπτωση η δική μου πρόταση είναι να φύγει αυτό το πράγμα, να μην υπάρχει τέτοια εξαίρεση, γιατί νομίζω ότι εκεί συμπυκνώνεται η μεγαλύτερη κίνδυνη κατά την άποψή μου. Ε, ευχαριστώ, δεν θα έχω τίποτα άλλο. Περιμένω να μου πείτε, να συνονιθούμε πότε πρέπει να καταθέσω το γραπτό κείμενο, να γίνει μετάφραση, να συνεχίσουμε την κουβέντα μας πιο, πιο συγκεκριμένα. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Χουντή ε, και ε, θα υπάρξει επαφή με τη γραμματεία, θα σας ενημερώσει η γραμματεία. Εν πάση περιπτώσει, εμείς και την επόμενη φορά ε, το βάζουμε το θέμα στην ημερήσια διάταξη και θα σας ε, πούμε και τον ε, χρόνο κατά την ημερομηνία κατάθεσης των τροπολογιών για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε τον Ιούνιο στην Ολομέλεια. Ιούνιο. Δεύτερο ήμις του Ιουνίου. Δεν ξέρω αν τελικά κάποιος να λάβει το λόγο. να έχω στείλει το κείμενο, με συγχωρείτε που είμαι λίγο σχολαστικό, αλλά να είμαστε σαφεί. Πρέπει να έχει σταλεί κείμενο για, την τρίτη, για τη συζήτηση στι 20 Μαρτίου. Αυτό εννοείται. Ναι, πείτε μου συγκεκριμένα, έτσι πρέπει να είναι. Μάλιστα. Πολύ σωστά κύριε Χουντή, μέχρι τις 20, ε, μάλλον στις 20 Μαρτίου, δηλαδή να σας το πω, για τις 20 Μαρτίου προβλέπεται η συζήτηση για το γραπτό σχέδιο που θα το παρουσιάσετε εσείς εδώ, εδώ να έρθετε 20 Μαρτίου και να το παρουσιάσετε. Πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο θέμα της ε, ημερήσιας ε, διάταξη 134 του 12 Ανέ Βερντιέ και Νατάσα Σικότη και είναι εδώ παρούσες ε, οι δύο υπογράφουσες που ε, υπογράφηκε και από άλλους 14 ε, πολίτες. Η κυρία Μπερτιέ ζήτησε το λόγο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο κυρία Μπερτιέ. Thank you. Ευχαριστώ. Η αναφορά δεν υπογράφτηκε από 60 πολίτες, αλλά από 60 μήκη όμικρον. Έχει πέντε σημεία λοιπόν η αναφορά ότι έχει αποτύχει η Κομισιόν να λύσει το πρόβλημα, το αίτημά μας για πληροφόρηση ούτε σεβάστηκε το χρονοδιάγραμμα που είχε προβλεφθεί για τις απαντήσεις. Ούτε σεβάστηκε τη σύμβαση, τη σχετική σύμβαση και την ούτε χορήγησε επαρκή πληροφόρηση για το περιβάλλον, ούτε μπόρεσε να αποδείξει ότι υπάρχει επαρκής και αποχρόν λόγος για την κατακράτηση της πληροφόρησης. Άρα παραβίασε και ορισμένες αποφάσεις του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητού. Πρώτον, τα απευθύναμε όλα στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος που έχει έναν εκπρόσωπο αν δεν απατώμε σήμερα εδώ και σε άλλες γουδού ενέργεια, μεταφορές, κλιματολογικές αλλαγές κτλ. Λοιπόν, πρώτον ότι δεν σεβάστηκε την υποχρέωση να συντάξει ένα μητρό ή δελτίο πληροφόρησης. Μελέτες, επιστημονικές μελέτες, τα συμπαράσματά τους για τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρουν τα κράτη-μέλη την ε, περιβαλλοντολογική ναμαθεσία. Δεν μας χορήγησε τα σχετικά έγγραφα ούτε για τις εκπομπές διοξιδίου και τις επιπτώσεις τους ως προς την βιομάζα. Δεν είχαμε καμία πρόσβαση. Η Κομισιόν απάντησε ότι υπάρχει απλή υποχρέωση ηλεκτρονικώς να χορηγούνται ορισμένα δεδομένα αλλά όχι λεπτομερή μητρώα. Αυτές όμως οι ηλεκτρονικές τράπεζες δεδομένων πρέπει να χορηγούν και πρόσβαση στο κοινό. Στο κοινό. Και όμως δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ούτε είναι σαφής η διαφορά που καθορίζει η Κομισιόν μεταξύ ηλεκτρονικής τραπέζης δεδομένων και διαθεσίμου μητρώου πληροφόρησης. Ο σκοπός πάντως ούτως ή άλλως είναι η χορήγηση της πληροφόρησης και δεν το σεβάστηκε αυτό, δεν έχει πρόσβαση, δεν χορηγεί πρόσβαση γιατί τη σχετική πληροφόρηση δεν την κατακρατεί μόνο η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος αλλά και Ενεργείας. Οι πολίτες που δεν γνωρίζουν τις λεπτομέρειες για τη λειτουργία της Κομισιόν δεν μπορούν εύκολα να βρουν αυτές τις πληροφορίες. Παράδειγμα, which provides really clearly that οι σχετικές οδηγίες προτυλέπουν την εύκολη πρόσβαση γιατί τα επίσημα αυτά έγγραφα είναι υποχρεωτικό να είναι διαθέσιμα. Πρέπει να εμφαίνονται σε κάποιο δημόσιο μητρό και δεν συμβαίνει αυτό ας πούμε στις συνεδριάσεις των τριμερών διαλόγων τα πρακτικά τους δεν χορηγούνται στο κοινό. Και άρα δεν μπορεί η κοινωνία των πολιτών να γνωρίζει πώς γίνεται, πώς ε, αποφασίζεται η κοινοτική ναμαθεσία. πολλές επιστολές ενδιαφερομένων που προσπαθούν να επηρεάσουν τους νομοθέτες και, αυτά πρέπει, και αυτές πρέπει να γίνονται γνωστές. Για να μειωθεί ο φόρτος εργασίας των υπαλλήλων της Κομισιόν θα έπρεπε ακριβώς το αντίθετο να γίνεται ή να χορηγούνται τα έγγραφα. Η να χορηγουνται τα εγραφα Ήρης ή της Ήριδος προβλέπει τέτοια πρόσβαση και όμως δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα η Κομισιόν. Αντίθετα προβλέπονται παράνομα εξαιρέσεις από τη χορήγηση αυτών των στοιχείων και κρατούνται ως απόρριτα επαναλαμβάνω σε παραβίαση της συνθήκης Ήρης. Επανειλημμένα η Κομισιόν μας αρνήθηκε πρόσβαση και τη ζητούμε και αυτή τη φορά με την ευκαιρία της αναθεώρησης της ε, συμβάσεως Ήρης να διευρύνει τη χορήγηση των, της πληροφόρησης και για την κοινωνία των πολιτών. Τέλος, δεν σεβάστηκε τα χρονικά όρια που προβλέπονται για την απάντηση, για τις απαντήσεις. Έχει γίνει πια συστηματικό αυτό το πρόβλημα να παραβιάζονται τα χρονικά όρια που προβλέπονται. Μία φορά μάλιστα και για δεύτερη φορά εξέπνευσε η διορία χωρίς απάντηση. η προβλεπόμενη φράση είναι όσο το δυνατόν συντομότερα, αλλά καμιά φορά αυτό σημαίνει μήνες ολόκληρους ή και χρόνια. Αυτό είναι απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Uh, with the and... Επανειλημμένα στείλαμε επιστολάς, δεν μας απάντησαν, τις ξαναστήλαμε και δεν μας ξανααπάντησαν. Αποτέλεσμα, η Κομισιόν αποκλείει από τους πολίτες, παραβιάζει το δικαίωμα των πολιτών στην πληροφόρηση και αυτό σε κατάφορη παραβίαση των συνθήκων που προβλέπουν διαφάνεια. Ευχαριστούμε Μπρέγκλαντ από την Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, είμαι εδώ με τον συνάδελφό μου δεν συμφωνούμε με την νομική ερμηνεία που έκανε η αναφέρουσα. Ε, δεν προβλέπεται τίποτε από όλα αυτά. Κάνουμε ακριβώς ό,τι προβλέπουν οι συμφωνίες. Οι επιστημονικές μελέτες αναρτώνται στην, ιστοσελίδα, στην αρμόδια ιστοσελίδα. Υπάρχουν βέβαια ορισμένες εκκρεμότητες, α, γιατί εκδικάζονται ορισμένες υποθέσεις στο δικαστήριο γι' αυτό. Τα νομοθετικά έγγραφα, η έλλειψη πληροφόρησης για τους τριμερείς διαλόγους, αυτό ισχύει και για το Κοινοβούλιο, όχι μόνο για μας όσο δε για το κύριο επιχείρημα την παραβίαση της σύμβασης Ντόρους, αυτήν που έλεγε η Ήρηση η προηγούμενη αναφέρουσα, εγώ δεν παρατήρησα καμία παραβίαση, το δικαστήριο επίσης δεν παρατήρησε καμιά τέτοια παραβίαση. Και όπως γνωρίζετε, ο κανονισμός όρος λέει αυτή τη φορά ο μιλητής καθώς και η 1367, ο κανονισμός 1367 που από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο δεν προβλέπουν τίποτε το παράνομο. Πού να φανταστεί κανείς τέτοιο πράγμα. Δεν τολμώ ούτε να το διανοηθώ. Όσο για τον κανονισμό 1367, δεν ξέρω αν θέλει εδώ ο συνάδελφός μου να προσθέσει τίποτα. Είπατε ότι η λύση που δώσαμε για την πρόσβαση στην περιβαλλοντολογική πληροφόρηση περνάει από το Γενικό Κανονισμό των 1049 δηλαδή, αλλά αυτό κάνει και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Υπάρχει σίγουρα τρόπος να βελτιωθεί η διαφάνεια. Εδώ συμφωνώ με τους αναφέροντες για περισσότερη διαφάνεια. Η γενική μου διεύθυνση προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί. Ό,τι μπορεί. Παραδείγματος χάρη στο εξή τις προειδοποιήσεις τις δημοσιεύουμε. Και για τα παράπονα των αναφερόντων Νομίζω ότι αυτά ξεπερνούν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Αυτό βέβαια δεν αποκλείει βελτίωση, αλλά προς τη στιγμή ξεπερνούν. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρος. Κυρία Όκεν. Με συντομία από ό,τι βλέπουμε μας είπατε ότι μπορείτε να καλύψετε δύο από τις πέντε αξιώσεις. Το θέμα είναι εάν θεωρείτε ότι είναι επικουρικού χαρακτήρα η σύμβαση του Άρχου σε σχέση με την υπόλοιπη νομοθεσία. Όμως, συνήθως κατησχύει η διάταξη, η νομοθεσία του διεθνού δικαίου. Ε, μα είπατε ότι είστε εδώ με την ιδιότητά σα ω υπαλλήλου και το σέβομαι αυτό. Όμω, είναι πάρα πολύ καλά τεκμηριωμένη και προετοιμασμένη αυτή η αναφορά. Έχει βάσιμα επιχειρήματα, είναι διατυπωμένη ξεκάθαρα. Οπότε, σεβαστείτε και εσείς τη δουλειά των αναφερόντων. Μην λέτε κάναμε ό,τι μπορούσαμε και ίσως το ένα ίσως το άλλο. Δεν νομίζω ότι αυτός είναι τρόπος να αντιμετωπίζει κανείς μια αναφορά με τη συνθήκη του Άρχους. Και επίσης είπαμε και για την αναθεώρηση της οδηγίας της ε, Επιτροπής Δομικής Ενέργειας. Και άλλωστε λέμε για το δικαστήριο. Μα περιμένουμε το δικαστήριο. Περιμένουμε η κομισιόν να επικαλεστεί τη συνθήκη του Άρχου, να τη χρησιμοποιήσει κλπ. Πάντα δίνουμε μάχη. Να υπάρχει διαφάνεια, να είναι οι πόρτες ανοιχτέ στον πολίτη και η Κομισιόν θα πρέπει επίσης να είναι πρωτοπόρος σε σχέση με τις και όχι να αποτελεί την τροχοπέδη για αυτές τις εξελίξεις. Άρα, για άλλη μια φορά, ας πούμε στην Κομισιόν, κάντε τη δουλειά σας, διαβάστε καλύτερα, μελετήστε την αναφορά και τα επιχειρήματα και απαντήστε στα όσα ξεκάθαρα εκεί τίθενται. Κύριε Κάσμα και το λόγο, σας ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, συγχαρητήρια προς τους αναφέροντας, διότι πάρα πολύ καλά τα λένε. Επίσης, ε, και εγώ συμμερίζομαι τον προβληματισμό, τις ανησυχίες και νομίζω ότι ξεκάθαρα πρόκειται από τα όσα είπε η Κομισιόν ότι εδώ έχουμε κατάφορη, κατάφορη παραβίαση της υποχρέωσης σεβασμού του, του πολίτη. Τα τρία θεσμικά όργανα είναι υπόλογα. Πού είναι οι νομοθετικές προτάσεις που θα πρέπει να κατεβάσετε. Γιατί εσείς προτείνετε νομοθεσία και οι υπόλοιποι συνομοθέτες ε, θεσπίζουν τη νομοθεσία και ενεργούν. Οπότε ακριβώς για το 1049 δεν αποδέχομαι αυτό το οποίο είπατε. Θα πρέπει έστω και με ένα θεώρηση να γίνει κάτι. Αλλά και το πιο σωστό είναι να προκάνετε κάποιες νομοθετικές προτάσεις που δεν θα έρχονται σε αντίφαση με τη του αρχού. Τώρα όσον αφορά τις προθεσμίες, οι προθεσμίες δεν είναι αυθαίρετες. Προέγυψαν από διαπραγματεύσεις με Κομισιόν και Κοινοβούλιο. Κατόπιν του Μαΐου του 2001, οπότε και θεσπίστηκε το 1049. Και τώρα, σε σχέση με το θέμα του στάθμισης του δημοσίου συμφέροντος. Πάρα πολύ σημαντικό είναι. Και γι' αυτό και όλα αυτά είναι πάρα πολύ βασικά η συνθήκη δηλαδή του Άμστερνταμ και της Λισαβόνας. Πώς λοιπόν θα έρθει πιο κοντά ο πολίτης στο ευρωπαϊκό όραμα. Και αυτό να γίνει τώρα. Τώρα που ο κόσμος αποστασιοποιείται, κρυώνει, απομακρύνεται όλο ένα και περισσότερο το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να κάνει την πορεία ούτως ώστε να πάμε για αναθεώρηση του 1049. Και το ξαναλέω, η Κομισιόν έχει γίνει το, το, το, το, το φρένο ή τροχοπέδι για να υπάρξει εξέλιξη κατόπιν εργασία Κοινοβουλίου και Κοινοβουλίου. Είναι παράδεικτο αυτό. Μα είναι δυνατόν να έχουμε τέτοια αντιμετώπιση ε, που να μην είναι περιπτωσιολογική, που να είναι γενική. Να τα, να τα καλύπτει όλα για το περιβάλλον, για τον για τέτοια σοβαρά πράγματα. Τέλο πάντων, είχα και εγώ κάποιε ερωτήσει για την Κομισιόν και του εκπροσώπου, αλλά τελικά ε, δεν τι ε, βάλω τι ερωτήσει για να αξίζει τον τρόπο. Γιατί άκουσα τι είπαν. Τέλο πάντων, εγώ έχω να σα ε, πω, σε εσά του ότι σε πρώτη ανάγνωση είχαμε συμφωνήσει, κάναμε ό,τι έπρεπε και αυτό το οποίο θέλουμε δεν είναι το να σας περιστύλουμε τα δικαιώματα αυτά τα οποία κατοχυρώνεται το 1049 κάθετος του 2001. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να εξασφαλίσουμε το ότι θα υπάρξει κάποιο είδου αναβάθμιση, αναβάπτιση αυτών των δικαιωμάτων. Και να, έχουμε νομολογία, να, να βεβαιώσουμε τους ε, Ευρωπαίους ότι δεν θα πρέπει να περιμένουν απόφαση του δικαστηρίου και τότε να απαντάει, τότε να κάνει κάτι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τελικά να, να, να, να, να κάνει αυτό που την υποχρεώνει το γεγονό ότι είναι υπόλογη στους πολίτες. Επομένως, εμείς είπαμε ότι θα πρέπει ο 1049 να ισχύει με κάθε επιφύλαξη όσον αφορά ε, τα όσα ε, ορίζει η σύμβαση του άρχους και θα πρέπει επομένως να ισχύουν τα όσα δικαιούται ο πολιτή όποτε θέλει να έχει πρόσβαση σε κάποια έγγραφα, γιατί τελικά αυτό καταντάει σχεδόν καυκικό. Όταν έχουμε κάποια βάση δεδομένων, στην οποία να έχει πρόσβαση το κοινό. Να υπάρχει, υποτίθεται έχουν πρόσβαση αλλά τελικά όταν έρχεται η ώρα να πάει κανείς να τα κοιτάξει, κάποιος να λέει όχι, δεν είναι για, το, για τον κόσμο αυτή η βάση δεδομένων. Εμείς θα πρέπει να είμαστε ε, ξεκάθαροι. Τι βάσει δεδομένων υπάρχουν, σε ποιον είναι προσβάσιμες κλπ. Εάν δεν είναι προσβάσιμες στο κοινό, είναι, τελείωσε. Είναι ανοιχτή, δημόσια. Και αν ε, δείτε τι γίνεται, ε, ε, αυτό είναι και τα, τα μητρώα, τα πρωτόκολλα. Τα, τα αγγλικά είναι η μητρική μου γλώσσα. Ξέρω τι είπα να πει. Ανοιχτή στο κοινό, ανοιχτή στον κόσμο, δημόσιο βάσει δεδομένων. Αυτό είναι αίτημα, απέτηση του, του, του πολίτη, των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Φυσικά και μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση εμεί ω κοινοβούλιο. Ναι. μπορούμε να συμφωνήσουμε. Και έτσι να εξασφαλίσουμε ότι τα έγγραφα είναι ανοιχτά, είναι διαθέσιμα. Αν μπορείτε απαντήστε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και Άουκεν, θέλετε ξανά το λόγο. Έχετε το λόγο. Ο, ο άλλος κύριος. Θα σας μιλήσω στα γερμανικά. Και θα είμαι σύντομος. Συμφωνώ και με όσου μίλησαν, όσοι στην δική μου θυμάμαι και με τον κύριο Κάσμα. Και τέλο πάντων θα πρέπει να δούμε ότι οπότε είναι θέμα ενημέρωση πληροφοριών. Ε, δεν θα πρέπει να θεωρούμε ότι κακόπιστα ενεργεί ο πολίτη και ότι απλώ το κάνει για να ενοχλήσει τον, τον υπάλληλο. Ε, πρόκειται για νομικά κατοχυρωμένο δικαίωμα. Πρόκειται για κάτι πάρα πολύ βασικό. Για το, το, το, το δικαίωμα πρόσβαση στα έγγραφα. Εάν δεν κάνουμε κάτι, τότε ε, ο κόσμος θα δεσπιστεί μαζί μας. Θα πρέπει να έχουμε μια ε, ισορροπημένη αντιμετώπιση. Προσοχή, γιατί είναι ε, όλοι, όλοι οι εμπλεκόμενοι να έχουν την ίδια πρόσβαση ας πούμε να μην, δίνουμε, μην αποκαλύπτουμε περισσότερα στη βιομηχανία από ότι στον πολίτη ή στην μη κυβερνητική οργάνωση. Οπότε και εμείς θέλουμε να κατοχυρώσουμε έτσι τον ακρογωνίο ρήθο της δημοκρατίας στη διαφάνεια. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίσει ε, με, τόση αποφασιστικότητα να, να, να, να μπλοκάρει αυτού του είδους την προσβασιμότητα με αυτές τις ε, τεχνητές διακρίσεις μεταξύ του το, το, πόσο ορίζεται το δημόσιο συμφέρον, θα πρέπει να υπάρχει κάποιο είδου μητρό, το οποίο να, να περιβάλλεται από εγγυήσει ελεύθερης πρόσβαση για τι πληροφορίε που περιέχονται εκεί. είναι δυνατόν να θεωρείται κάτι εμπιστευτική πληροφορία όταν κάποιο υποβάλλει κάποιο αίτημα εξέτασή τη και μετά αρχίζουν τι καθυστερήσει και αυτά. Έχουμε δικαιολογημένη απέτηση πρόσβαση στην πληροφορία. Και η Κομισιόν προσπαθεί να παρελκύσει τις εξελίξεις αντί να ανταποκριθεί. Είναι σαν να κορυδεύεται τον κόσμο υπονομεύεται τη δημοκρατία, τη διαφάνεια. Θεωρώ ότι είναι υποχρέωση, η ιερή μας υποχρέωση να επιβάλλουμε στην ε, Επιτροπή να αλλάξει νοοτροπία, να συμμορφωθεί με την σύμβαση του άρχους και να σταματήσουν ε, αυτά, αυτά τα παραδείγματα της κατάφορης κακοδίκησης. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιο άλλο το λόγο ή αν ε, θέλετε από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβετε το λόγο για να απαντήσετε. Έχει το λόγο, κύριε Πληγό. Όχι να αρχίσουμε πολιτική συζήτηση, αλλά να δούμε το πώς μπορούμε να καλύψουμε ε, την, ε, τα όσα είπαν οι Έχουμε 6.000 αιτήματα Ε, παροχής πληροφοριών και απορρίπτουμε 80 από αυτές. Πολύ, πολύ μικρό είναι το ποσοστό ε, του όχι που λέμε. Θα πρέπει να ε, διαπιστώσουμε ότι είναι Σημαντικό αυτό που λένε αναφέροντα, αλλά θα πρέπει να το δούμε για πιο πέρα το θέμα και θα πρέπει να δούμε το ότι υπάρχει εδώ πέρα κάποια ε, δυσκολία και όπω η κυρία Άουκεν θα πρέπει να πούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αρχίσει να ενεργεί συμμορφούμενη προς την νομοθεσία. Γιατί άλλωστε και ενώπιον της Επιτροπής Λίβεως και ο κύριος ε, Κάσμαν εξετάζεται αυτή η αναθεώρηση της νομοθεσίας. Και εμείς θα πρέπει, με αφορμή τα όσα ελέγχθησαν σήμερα εδώ, να γράψουμε στην Τροπή και να συνεργαστούμε μαζί της, ούτως ώστε να υποστηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Και έτσι να καλύψουμε και το αίτημα των αναφέροντων. Κύριε Κάσμα, έχετε το λόγο. Θα είμαι σύντομος. Και ως εισηγητής της έκθεσης για την αναθεώρηση του κανονισμού, ευχαρίστως να ζητήσω από την Επιτροπή Λίμπε να λάβει υπόψη αυτή την αναφορά, άρα θα πρέπει να μείνει ανοιχτή, είτε μέχρι ότου ικανοποιηθεί το αίτημα, είτε μέχρι ότου ολοκληρωθεί η αναθεώρηση της νομοθεσίας. Βέβαια, λέει ο Πρόεδρος. Νομίζω λοιπόν ότι η ε, αναφορά αυτή παραμένει ανοιχτή και θα συνεργαστούμε και με την ε, Επιτροπή ΛΥΜΠΕ η οποία ασχολείται με την οδηγία για την πρόσβαση στα έγγραφα. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή, ευχαριστώ τις υπογράφου για τη συμμετοχή ε, στη συζήτηση και προφανώς θα ξανασυντούμε για να δούμε πώς θα προχωρήσει αυτή η συγκεκριμένη αναφορά. Σας ευχαριστούμε πολύ και πάμε τώρα στο επόμενο θέμα που είναι η επόμενη αναφορά Γιάν Φλόρι θα μας παρουσιάσει την ε, αναφορά. Πέντε λεπτά έχετε στη διάθεσή σας. Ε, δίνω το λόγο ε, στον πρώτο υπογράφουσα αυτής της αναφοράς. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτέ, ευχαριστούμε για την πρόσκλησή σας. Με την Στέφανο Σιανίκ που είναι πρώην ανθρακορίχος εκπροσωπούμε την οργάνωση Ντεστό Καμίν. Έχουμε και διαφάνειες. Βρισκόμαστε στο Βίτελσχάιμ στην Αλσατία και ενδιαφερόμαστε για ένα υπόγειο απόθεμα ύδατος όπου έχουν εναποτεθεί τοξικά απόβλητα θεωρούμε ότι είναι ανυπεύθυνο και ότι παραβιάζει τις ευρωπαϊκές οδηγίες, ε, οδηγίες αυτή η μόλυνση. Εδώ βλέπετε το πρόβλημα εκτός από τους διερμηνείς. Τα τοξικά αποθέματα είναι δίπλα στο ρήνο και ο χώρος απόθεσης βρίσκεται 550 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, κάτω και από την ε, υδατική εναπόθεση. Αλλά φτάνει μέχρι εκεί. Τα απόβλητα κατεβάστηκαν από αυτήν τη σύραγγα Η άδεια χορηγήθηκε το 1997 και άρχισε η αναπόθεση το 1999. Το 2002 σημειώθηκε μια πυρκαγιά και σταμάτησε η χρήση του ορυχείου. Η πυρκαγιά οφειλόταν στα απόβλητα που βρίσκονταν σε σάκους όπου έγραφε αμίαντος. Αλλά δεν έχει ελεγχθεί αυτό. Το 2010 εμφανίστηκαν δύο εκθέσεις του Μάρκο Καφέ και της οργάνωσης Ντρεάλ Αλσαρτίας και μετά μια τοπικής επιτροπής εποπτείας. Αυτές οι τρεις εκθέσεις έχουν την, τα ίδια συμπεράσματα. Εδώ βλέπετε εκτός από τους μισούς διερμηνείς λοιπόν πώς έχουν τα πράγματα. Έχουν τα ίδια συμπεράσματα λοιπόν οι τρεις εκθέσεις. Πρώτον, ότι δεν μπορεί να αποφευχθεί η μόλυνση και του ορυχείου ότι η μολυσμένη σαλαμούρα θα ανέλθει και στην επιφάνεια και θα μολύνει και το πόσιμο είδωρ. Είναι σαφές αυτό. Και η έκθεση της Κοπίλ βεβαιώνει ότι θα υπάρξει και μόλυνση από υδράργυρο. Τονίζει επίσης ότι και άλλοι ρήποι όπως το αντιμόνιο, το αρσενικό και άλλα βαρέα μέταλλα θα μολύνουν. Η έκθεση αναφέρει ότι το βούλωμα των ε, σειράγκων με μπεντονίτη δεν θα αρκέσει και δεν υπάρχει καμία εγγύηση μακροπρόθεσμα ότι θα αποφευχθεί η μόλυνση που τελικά φαίνεται ότι είναι αναπόφευκτη. Ποια είναι η θέση του γαλλικού κράτους. Η άδεια που δόθηκε για την αναπόθεση των αποβλήτων εξαιρεί μόνο την περίπτωση σοβαρού ατυχήματος. Αλλά αυτό υπήρξε το 2002, η πυρκαγιά. Το 2012 το κράτος αποφάσισε να μεταφέρει αλλού ορισμένα από αυτά τα απόβλητα. Χρειάστηκαν όμως 10 χρόνια και 55 εκατομμύρια ευρώ δημοσίου χρήματος για να δεχτεί το κράτος να εξετάσει τα πράγματα. Γιατί τέτοια καθυστέρηση ορισμένοι θέτουν το ερώτημα και αναρωτιούνται μήπως υπάρχει κάτι τώρα διενεργό στα μεταξύ των αποβλήτων. Η απομάκρυνση των ε, καταλήπων ε, ε, δεν βοηθάει βέβαια την ποιότητα του πόσιμου νερού η απομάκρυνση των καταλήπων λοιπόν, υδράργυρου. Αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει, ε, διότι υπάρχουν ολόκληρα μπλοκ από υδράργυρο και πώς μπορεί κανείς ε, να επιτύχει αυτή την απομάκρυνση. Ε, δεν είναι εύκολο να γίνει αυτή η απομάκρυνση. Ένας ε, ελβετός ε, εμπειρογνώμονας ε, κατέληξε στο ότι είναι πολύ πιο εύκολο να υπάρξει απομάκρυνση όλων των αποβλήτων χωρίς να δαπανηθούν περισσότερα χρήματα. Το θέμα είναι ότι όσο περισσότερο καθυστερούμε, τόσο πιο δύσκολο είναι να απομακρυνθούν απόβλητα. Αξιότιμοι πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτέ, ε, καλούμε το γαλλικό κράτος να αναθεωρήσει τη στάση του, γιατί θεωρούμε ότι είναι υποχρέωσή του να ε, μεριμνήσει για το μέλλον των μελλοντικών γενεών και να τηρεί τις ε, ε, διατάξεις της οδηγίας ε, επικαλούμενο το, επικαλούμενη το άρθρο 147 που λέει ότι πρέπει να προστατεύουμε το περιβάλλον με βάση την αρχή της αποφυγής και της πρόληψης. Όχι, θέλω να προσθέσω ότι ήμουν ανθρακορίχος και επί 32 χρόνια και γνωρίζω ακριβώς, σε αυτό το ρηχείο και γνωρίζω ακριβώς το πρόβλημα. Είναι πολύ απλό. Ή θα αφήσουμε τα απόβλητα ή θα τα βγάλουμε. Και αν τα αφήσουμε τότε είναι απολύτως βέβαιο ότι τα παιδιά μας θα μας πούνε μετά ότι τα δηλητηριάσαμε. Ενώ άμα τα μεταφέρουμε ε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μία είναι λοιπόν η λύση όλα αυτά τα απόβλητα να αποσυρθούν. Και γίνεται, είναι δυνατόν. Και όσο καθυστερούμε τόσο χειρότα γιατί υπάρχει η διαρροή τους. Ο κύριος Ορμπάν. Σας κατευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η έλαβε πληροφόρηση για αυτή την αναφορά το 2012. Την εξετάσαμε αυτή την πληροφόρηση και διαπιστώσαμε ότι το πρόβλημα συνδέεται με την οδηγία εναπόθεσης ή χωματερών που προβλέπει ορισμένα κριτήρια για την αδειοδότηση και την εποπτεία. Η τελική απόφαση με βάση αυτά τα κριτήρια θα ληφθεί από τα κράτη-μέλη όμως και δεν βρήκαμε χρόνο ακόμη. Δεν βρήκαμε καμία απόδειξη ότι δεν τηρούνται από τις γαλλικές αρχές τα κριτήρια. Και η οδηγία για τα υπόγεια ύδατα που αναφέρει εδώ αναφέρον απαιτεί από τα κράτη-μέλη να αξιολογήσουν τη χημική σύνθεση των υπογείων υδάτων για να διαβεβαιώνεται η μη μόλυνσή τους. Μέχρι το 2015 απαιτείται αυτό. Οι δε γαλλικές αρχές το έπραξαν αυτό γιατί μέχρι τώρα εφάρμοσαν τα σχέδια ελέγχου των υπογείων υδάτων και έλαβαν τα μέτρα που έπρεπε ώστε τα υπόγεια ύδατα να καθαριστούν μέχρι το 2015. Άρα δεν βρίσκουμε τίποτα που να λέει ότι οι γαλλικές αρχές παραβιάζουν τις οδηγίες. Τότε επίσης Μία από τις τρεις εκθέσεις που αναφέρονται την είδαμε και αυτή δείχνει ότι οι γαλλικές αρχές γνωρίζουν τα προβλήματα στον τόπο εκείνο και άρα είναι και διατεθειμένες να βρουν, να εφαρμόσουν μία αποδεκτή λύση. Τώρα είδα από την παρουσίαση εδώ ότι υπάρχουν και νέα στοιχεία διότι οι αναφέροντες μίλησαν για μία έρευνα ελβετών εμπειρογνωμόνων στα τέλη του 12 και είπαν ότι υπήρξε μια απόφαση μερικής απομάκρυνσης των αποβλήτων άρα μπορώ να πω ότι όταν θα έχουμε τη σχετική πληροφόρηση θα την αξιολογήσουμε δεόντως. Αλλά πρέπει να έχουμε τις λεπτομέρειες που δεν τις γνωρίζαμε. Όταν. Ευχαριστώ. Μιλιέ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε μου. Ευχαριστώ και τους αναφέροντες και τις αναφέρουσες για την παρουσία τους και την σαφή τους πληροφόρηση. Θα ήθελα να επανέλθω σε ένα αριθμό στοιχείων, νέων στοιχείων, ως προς τουλάχιστον σύμφωνα με, σε σύγκριση με τα αποτελέσματα του περασμένου Νοεμβρίου της Κομισιόν. Χαίρομαι ιδιαίτερα που αναγνωρίζει ότι υπάρχουν νέα στοιχεία, βάσει των οποίων παραμένει το πρόβλημα εκεί και δεν έχει λυθεί τίποτα. Δεν σας κρύβω ότι ξέρω πολύ καλά τα πράγματα της περίπτωσης αυτής, γιατί πριν από 15 χρόνια το πρώτο θέμα που χρειάστηκε ως δικηγόρος στην Αλσατία να χειριστώ ήταν αυτό. Γιατί μόλι άρχισε να λειτουργεί αυτή η χωματερή, η εναπόθεση επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων, τέθηκαν και τα προβλήματα από τότε μέχρι σήμερα. 15 χρόνια αργότερα λοιπόν ο κίνδυνος παραμένει ακέραιος και αν δεν δοθεί ικανοποιητική απάντηση από το γαλλικό κράτος τότε οι αλσατικές αρχές θα απευθυνθούν στους ευρωβουλευτάς. υπόθηκε ότι 44.000 τόνοι τοξικών αποβλήτων έχουν εναποτεθεί εκεί σε βάθος μεγαλύτερο των 500 μέτρων κάτω από υπόγεια ύδατα που είναι η μεγαλύτερη υπόγεια πηγή ποσίμου ύδατο στην Ευρώπη και υπάρχει αποδεδειγμένος κίνδυνος μόλυνσης τους και αυτό θα αφορά την υγεία πολλών εκατομμυρίων Ευρωπαίων. Το μόνο, η μόνη αποδεκτή λύση όπως είπαν και οι αναφέροντες είναι οι γαλλικές αρχές να ανταποκριθούν στην υποχρέωση που έχουν για την προστασία να μεταφέρουν πλήρως όλα τα τοξικά εκεί απόβλητα αλλού. Προς στιγμή, ενώ εδώ και 10 χρόνια δεν λειτουργεί η χωματερή, δεν έχει γίνει τίποτα για την απομάκρυνση. Απλώς βουλώνουν ορισμένες σύραγγες και επιτηρείται λένε το υπόγειον είδωρ. Αλλά αυτό δεν είναι σοβαρό και αυτή η έλλειψη σοβαρότητας παρατηρείται εδώ και 15 χρόνια. Για 30 χρόνια προβλεπόταν η λειτουργία της χωματερής μετά από λιγότερα από πέντε χρόνια έκλεισε λόγω της πυρκαγιάς που είπαν οι αναφέροντες. Πυρκαγιάς που οφειλόταν στην εναπόθεση αυτών των τοξικών αποβλήτων. Σας υπενθυμίζω ότι εδώ μιλάμε για τοξικά βιομηχανικά απόβλητα, δηλαδή ράργυρο, κιάνιο, αρσενικό, αμίαντο κλπ. Η αρχική αδειοδότηση προέβλεπε τη μεταφορά το πολύ σε 30 χρόνια όλων αυτών των αποβλήτων ή μετά από σοβαρό ατύχημα. Σημειώθηκε το ατύχημα πριν από 10 χρόνια και δεν λήφθη καμία απόφαση. Μετά από τη σύσταση της Κομισιόν η Γαλλία δήλωσε ότι βάσει μελετών εμπειρογνωμόνων γνωρίζει το πρόβλημα και ότι είναι διατεθειμένη να σεβαστεί ό,τι προβλέπουν οι οδηγίες για τα απόβλητα, για τα υπόγεια ύδατα κτλ. Τον Δεκέμβριο του 12 έγινε αυτή η δήλωση και δεν είναι σωστή ανταπόκριση γιατί νομικά μεν η μερική μόνο απομάκρυνση των αποβλήτων δεν είναι ικανοποιητική και από την άλλη η απομάκρυνσή τους μπορεί να μην είναι και πολύ εύκολη. Γιατί είναι πολύ επικίνδυνη, θα ήταν πολύ επικίνδυνη και για τους εργαζόμενους που θα έκαναν αυτή τη μεταφορά. Je vais revenir, j'aurais vous évoquer les différents risques qu'on qu'on Λοιπόν, οι εμπειρογνώμονες ανέφεραν όλους τους πιθανούς κινδύνους και είπαν ότι είναι απαραίτητο να γίνει κάτι, αλλά χωρίς να επανέλθω τώρα σε όσα είπε ήδη Κομισιόν, Το γαλλικό κράτος προέβλεψε μια χρηματοδότηση 100 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά υπάρχει νέα εμπειρογνωμοσύνη από τον Ιανουάριο, ελβετική, του Μάρκου Μπούζερ, που είναι ειδικό για πυρηνικά απόβλητα και που έχει επιτυχώς μεταφέρει τέτοια απόβλητα και μας λέει ότι είναι δυνατή η απομάκρυνση και με κόστος το μισό από αυτό που προβλέφθηκε. Ερωτώ λοιπόν την Επιτροπή μας, καταρχήν ζητώ, να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά και να οργανωθεί επίσκεψη, διασταύρωση του Στοκαμίν στην Αλσατία και του Ελβετικού, της Ελβετικής χωματερής. Και ρωτώ γιατί ενώ τόσες μελέτες λένε ότι είναι επικίνδυνα τα πράγματα δεν γίνεται ολική απομάκρυνση. όλοι και οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες που γνωρίζουν τα θέματα της απομάκρυνσης των αποβλήτων λένε ότι είναι δυνατόν και με λιγότερο από 100.000 ευρώ. Γιατί λοιπόν το γαλλικό κράτος ενώ διαθέτει όλα αυτά τα στοιχεία δεν προτείνει παρά μόνο μερική απομάκρυνση και όχι ολική τη αυτή. Σας ευχαριστώ. κυρία Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε εκπρόσωποι της Κομισιόν. Θέλω να σας πω ως Ευρωβουλευτής από την Αλσατία ότι υποστηρίζω πλήρως αυτά που είπε η οργάνωση στο Καμίν και χαιρετίζω την παρουσία εδώ των δύο αναφερόντων. Η απάντηση όμως της Κομισιόν με απογοήτευσε. Βλέπετε και από, τα, από τις διαφάνειες που επιδείχθηκαν ότι η εναπόθεση τοξικών αποβλήτων στο πρώην ορυχείο άλατος μολύνει τα φρέατα, τα ύδατα, τα υπόγεια ύδατα που διασφαλίζουν το 50% του πόσιμου ύδατος ολόκληρης εκείνης της περιοχής από 44.000 τόνους πολύ επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων, υδράργυρο, αργενισενικό κλπ. Από το 1999 η αναπόθεση έγινε με περίεργο και επικίνδυνο τρόπο και εδώ και 11 χρόνια δεν γίνεται τίποτα. Επίσημες δε μελέτες έχουν αποδείξει ότι η επαφή μεταξύ υπογείων υδάτων και τέτοιων τόπων είναι κάτι ιδιαίτερα επικίνδυνο Όλες οι μελέτες δείχνουν ότι τα ύδατα εκεί έχουν ήδη αρχίσει να μπαίνουν στο παλιό ορυχείο και ότι θα υπάρξει πολύ πιθανή μόλυνση. Επίσης οι μελέτες δείχνουν ότι η ολική μεταφορά είναι δυνατή εφόσον έχουν ήδη ταυτιστεί και οι εναλλακτικοί τόποι εναπόθεσης. Επομένως είναι απαραίτητο και επίγον να γίνει η μεταφορά αυτή. Απογοητεύομαι πολύ λοιπόν από την ανεπαρκή απάντηση της Κομισιόν φαντάζομαι ότι θα την αναθεωρήσει. Αυτό είναι πολύ καλό παράδειγμα, υπόδειγμα σχεδόν ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας. Γιατί η Κομισιόν αγνοεί τους μελλοντικούς κινδύνους της μόλυνσης των ρινανίων υδάτων. Πρέπει να σκεφτούμε το μέλλον, το κοντινό μάλιστα μέλλον. Γιατί σε άλλους τόπους εναπόθεσης αντέδρασαν οι τοπικές αρχές με πλήρη απομάκρυνση των τοξικών αποθεμάτων. Είναι κάτι απολύτως δυνατόν, έχει ξαναγίνει. Όπως το Βίτελσχάιμ το ίδιο πρέπει να γίνει. Έχει χιλιάδες αναφέροντες και αναφέρουσες από όλα τα πολιτικά κόμματα συμφωνούν και πρέπει πολύ σύντομα να αναλάβουμε όλες τις ευθύνες μας και απαιτώ από το γαλλικό κράτος να σεβαστεί τις ευθύνες, να λάβει τις ευθύνες τους ευχαριστώ, του. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, σας, σας διαβεβαιώ. Μισό λεπτάκι θέλω. Τα έχουμε πει πολλές φορές, αλλά θέλω να υποστηρίξω τους ε, αναφέροντες. Και θέλω να επιβεβαιώσω αυτό το οποίο είπαν οι συνάδελφοι τόσο άρτια Υποστήριζω την αναφορά. Οπότε θα πρέπει να, το, να μην ανοιχτεί, να βαθύνουμε και η Κομισιόν δεν θα πρέπει να θεωρεί ότι αρκούν τα όσα κάνει η Γαλλία. Θα πρέπει να εξωθήσουμε σε, σε δράση περαιτέρω την Γαλλία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι υπάρχει απόλυτη συνένεση. Ελπίζω να ικανοποιήθηκαν και οι υπογράφοντες και νομίζω ότι τελικά όλοι συμφωνούν όσον αφορά στη συμπεριφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία υπολείπεται κατά πολύ από τον τρόπο που θα έπρεπε να συμπεριφερθεί ε, σε τέτοιου είδους ε, περιπτώσεις. Η Επιτροπή ε, Αναφορών νομίζω ότι πρέπει να κάνει πολλά περισσότερα και το πρώτο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να ξεκινήσει άμεσος διάλογος με τις ε, γαλλικές ε, αρχές. Να τις ε, ρωτήσουμε τι ακριβώς προτίθενται να κάνουν πολύ συγκεκριμένα πέρα από όλα αυτά που μας λένε με τις ανακοινώσεις τους, διότι από όσα ακούσαμε σήμερα και από όσα είδαμε, η κατάσταση που μεταξύ άλλων διαρκεί εδώ και 30 χρόνια δεν μπορεί πλέον να περιμένει άλλο. Είναι λοιπόν απολύτως απαραίτητο να υπάρξει κάποια παρέμβαση. Γι' αυτό λοιπόν ας δούμε τελικά τι θα κάνουμε και τι χρονοδιάγραμμα έχουν οι γαλλικές αρχές. Και μετά θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να μπει στην ουσία του θέματος και εμείς αναμφίβολα θα στηρίξουμε την όλη υπόθεση γιατί με τις πληροφορίες που θα συγκεντρώσουμε θα στηρίξουμε αυτή την έρευνα περιμένοντας λοιπόν να υπάρξει και μία απάντηση που θα είναι πιο κοντά ε, στις ε, ανάγκες των ε, πολιτών. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο άλλο. Ε, το τελευταίο σημείο της ε, διάταξη διάταξης θα το αναβάλουμε και ενημερώσαμε, ζητήσαμε και από τον εκπρόσωπο της Κομισιόν έρθει εδώ το απόγευμα. Έτσι λοιπόν, για να μην επιβαρύνουμε κυρίως ε, τους ε, διερμηνείς, κλείνουμε εδώ τώρα και θα ξαναξεκινήσουμε οι εργασίες μας το απόγευμα στις 3 ώρα. Γεια σας.